Καταρχάς, να σας καλωσορίσω μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές εδώ στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής Απασχόλησης. Ελπίζω να περάσατε ένα εξαιρετικό καλοκαίρι. Για μένα προσωπικά το καλοκαίρι ποτέ δεν φτάνει, αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Πρώτα λοιπόν ε, να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη χωρίς τροποποιήσεις. Παρακαλώ για την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Να σας ανακοινώσω επίσης ότι σήμερα έχουμε διαθέσιμες όλες τις γλώσσες του γλωσσικού μας προφίλ. Αν δεν υπάρχουν σχόλια ή παρατηρήσεις, μπορούμε επίσης να εγκρίνουμε και τα πρακτικά. Και έτσι πάμε στο Γενικό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Δημοσιονομικό έτος 2020, όλα τα τμήματα. Εγώ είμαι η υπεύθυνη εισηγήτρια. Απλώς να σας παρουσιάσω πολύ γρήγορα λοιπόν το σχέδιο της γνωμοδότησης που έχω συντάξει. Αυτό που τονίζω είναι την ε, προτεραιότητα στις ε, πολιτικές απασχόλησης και την απασχολησιμότητα. Νομίζω ότι ε, πρέπει να κοιτάμε τα αποτελέσματα και όχι το τι παράγει η χρήση των κονδυλίων, γιατί στην ουσία πρέπει να δούμε πόσο χρήσιμη είναι η χρήση των κονδυλίων, πόσο αποτελεσματική είναι η χρήση των κονδυλίων. Επίσης, έχω αναφέρει τις ε, τεράστιες προκλήσεις ε, που βρίσκονται μπροστά μας, όπως είναι η γύρανση του ευρωπαϊκού πολυπληθυσμού, οι δημογραφικές αλλαγές και γι' αυτό έχω αναφέρει και κάποιες προτεραιότητες που βλέπω, όπως είναι η κοινωνική ένταξη εκείνων που δεν έχουν δυνατότητα κοινωνικής ένταξης, άτομα με αναπηρία, κοινότητες όπως η Ρωμά σε κάποιες χώρες για παράδειγμα και οι γυραιότεροι, οι ηλικιωμένοι. Δεν έχουμε πια την πολυτέλεια να εξαιρούμε συγκεκριμένες κοινότητες από την ε, κοινωνία μας ε, γιατί θα τους χρειαστούμε για την εργασία. Αυτά από μένα για το σχέδιο γνωμοδότησης. Τώρα δίνω το λόγο στους σκιώδες εισηγητές για το ΕΛΚ, ο κύριος Τόμας ε, Τζεχόφσκι για τους σοσιαλιστές Μπράντο Μπενιφέ για το Ρινιού η κυρία Γιάννα Τούμ και για τους ε, πράσινους η Κατρίν Λάγκεν Ζίπεν. Δεν έχουμε στο ID ε, κάποιον εισηγητή ούτε στο ECR. Κύριε Ζεχόφσκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, να σας ε, συγχαρώ, γιατί σήμερα θα έχουμε την πρώτη ψηφοφορία για τη γνωμοδότησή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι πραγματικά για σας ε, ένα γεγονός που μάλλον αξίζει να εορταστεί. Θυμάμαι ε, τη χώρα σας. Ε, είχα πάει πριν από πέντε χρόνια. Είναι ένα πολύ καλό, ωραίο κράτος. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, για την ε, συνεργασία. Έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά εδώ και πολύ καιρό έτσι ώστε να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει ένα καινούριο στυλ, μια καινούρια, ένα καινούριο τρόπο εργασίας που δεν θα βασίζεται μόνο στις πλειοψηφίες αλλά στις συζητήσεις ε, και στην, στο βαθύ συλλογισμό. Σε αυτήν την γνωμοδότηση έχουμε όλους τους βασικούς τομείς. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό ε, να δούμε πώς θα εφαρμοστούν αποτελεσματικά τα κονδύλια που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του 2020. Δεν θέλουμε να υποστηρίξουμε προγράμματα που δεν έχουν νόημα και ξεκάθαρα αποτελέσματα. Θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένα συγκεκριμένο κέρδος ε, προγράμματα τα οποία θα φέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα ε, και ε, επίσης θα πρέπει να βασιστούμε στον αυτοματοποιησμό, στον αυτοματοποίηση, συγγνώμη. θα πρέπει να δούμε πώς τα διάφορα μέτρα και προγράμματα ε, θα οδηγήσουν ώστε να έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να κάνουμε νέα βήματα σε αυτούς τους νέους τομείς. Νομίζω ότι αυτά ήταν τα βασικά που ήθελα να τονίσω. Είμαι πεπισμένος ότι το σχέδιο προϋπολογισμού ε, θα πετύχει τους στόχους αυτούς. Τώρα το λόγο θα πάρει κύριος, η κυρία Χόμσε στη θέση του ε, Μπράντο Μπενιφέη. Ευχαριστώ. Θα πάρω το λόγο, αλλά έχω το κείμενο στα Ιταλικά. Θα το διαβάσω, αν δεν σας πειράζει, Ιταλικά. Είμαστε υπέρ του σχεδίου γνωμοδότησης και χαιρόμαστε πάρα πολύ που η συντάκτρα τη εκνομοδότηση ήδη από την γνωμοδότηση αυτή έχει θέσει κάποιε πρώτε προτεραιότητε που θα πρέπει να λάβει υπόψη τη η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή, Επιτροπή Προπολογισμών δηλαδή. Ω ομάδα σοσιαλιστών και δημοκρατών καταθέτουμε ορισμένε τροπολογίε οι οποίες θα πρέπει να συμπληρώσουν τις ήδη υποβληθήσεις δημοσιονομικές τροπολογίες τις οποίες έχουμε υποβάλει στο παρελθόν. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε τη συμβολή των κοινοτικών προγραμμάτων στον τομέα της απασχόλησης, ιδίως όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Επίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερο το πρόγραμμα ΕΑΖΗ για την απασχόληση και την κοινωνική κοινοτομία, καθώ επίση και όλα τα προγράμματα εκείνα, όπω το ΦΕΑΤ, που έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση τη ένδυα και του κοινωνικού αποκλεισμού. Για όλα αυτά τα προγράμματα είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε την κατάλληλη χρηματοδότηση, η οποία να προσαρμόζεται πραγματικά στι προκλήσει που καλούν τα ταμεία αυτά να αντιμετωπίσουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων να δαπανώνται με τον κατάλληλο τρόπο και να τηρούνται τα ανώτατα πρότυπα διαφάνειας κατά τη διαχείριση των ταμείων αυτών. Ιδίω θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να επενδύει στην πολιτική απασχόλησης για τους νέους, καθώς επίσης και για το ζήτημα της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των πιο νέων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί λοιπόν με τον συνάδελφο Μπενιφέη έχουμε υποβάλει τροπολογίες προκειμένου να αυξηθεί η χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερο την εγγύηση για τους νέους, ιδίω για τις χώρες εκείνες που πλήττονται από υψηλά επίπεδα ανεργίας. Τα 16 εκατομμύρια ευρώ προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επαρκούν. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αυξηθούν πολύ περισσότερο τα κονδύλια αυτά και ελπίσουμε ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι από τις άλλες πολιτικές ομάδες θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν αυτή μας την πρωτοβουλία. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα εξ της ομάδας Renew, το λόγο κυρία Γιάννα Τούμ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τόμ προφέρεται το επίθετό μου. Ενδεχομένως να μην γνωρίζετε ότι υπάρχει μια άλλη συνάδελφος που ονομάζεται Τούμ. Θα κάνω κάτι το δυνατόν προκειμένου να προφέρω σωστά το όνομά σας, λέει Πρόεδρος. Λοιπόν, Νομίζω ότι δεν μπορούμε να προσθέσουμε πάρα πολλά πράγματα. Δίδετε τη σωστή έμφαση στι σωστέ προτεραιότητε στο κείμενό σα. Όπω λέτε, όντω θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειε προκειμένου να ενσωματώσουμε όλε τι αποκλεισμένε κοινωνικέ ομάδε, τι ομάδε ΛΟΑΔΜΑ, και θα πρέπει προφανώς να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση υπάρχει κατά των ηλικιωμένων εργαζομένων. Τώρα για πέντε χρόνια στην Επιτροπή αυτή υπήρχε μια ευρύτερη συνένεση για τα ζητήματα αυτά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όμω να μπορούμε να λάβουμε υπόψη τις απόψεις όλων των πολιτικών ομάδων. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασκήσουμε πίεση στους συναδέλφους και από τις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές προκειμένου να καταφέρουμε μέσω του έργου μας, αυτού εδώ στην Επιτροπή Απασχόλησης, να βελτιώσουμε εν γέννη τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Πολύ συχνά στο παρελθόν έχουμε καταφέρει να πετύχουμε πολύ θετική πρόοδο στα πλαίσια τη συζήτηση που κάνουμε εδώ στην Επιτροπή μα και καταλήγουμε όμω τελικά με έναν κατάλογο ψηφοφοριών με πολλά αρνητικά πρόσημα σε πολύ σημαντικά για μα σημεία. Αυτό θα πρέπει προφανώ το αποφύγουμε στο μέλλον. Προσβλέπω λοιπόν σε μια επικοδομητική συνεργασία και είμαι πεπισμένη ότι μπορούμε να τα πάμε πολύ καλύτερα. Κυρία Τόμα, εγώ σα υπόσχομαι ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια και πρόφερα σωστά αυτή τη φορά το όνομά σα. Μπράβο, πολύ ωραία. Ας περάσουμε τώρα στους πρασίνους. Η κυρία Σίμπεν έχει το λόγο. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Αγαπητή Πρόεδρε, και εγώ έχω μερικά λόγια για εκ μέρου ε, των Πρασίνων. Χαίρομαι για μια πολύ καλή, επικοδομητική και αλληλέγγυα συνεργασία που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχουμε ανάγκη, ε, έχουμε τα εθνικά μας κράτη ε, και πρέπει να έχουμε μια κοινωνική Ευρώπη μαχόμαστε και μια κοινωνική Ευρώπη και αυτό πρέπει να αντικατοπρίζεται και εδώ. Για τα κοινωνικά project χρειάζονται χρήματα. Ε, ε, αυτά αποφασίζονται εδώ συζητούνται όπως και στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και πρέπει κανείς να τα υποστηρίζει γιατί χωρίς τα χρήματα δεν μπορούμε να έχουμε πολλά και σημαντικά ε, προγράμματα. Όπως θα δείτε για μας ε, η ανεργία των νέων ε, είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα δείτε στη λίστα ψηφοφοριών που μας ενδιαφέρει, ενδιαφέρουν. Όμως η ανεργία στην Νότια Ευρώπη τουλάχιστον 10 ε, χρόνια τώρα που υπήρχε η κρίση είναι κάτι που πλήττει τη νέα γενιά και δεν πρέπει να ξεχνούμε πόσοι νέοι άφησαν τη χώρα τους ε, για να, μπορέ... να φύγουν, ε, να πάνε σε μια άλλη χώρα όπου πρέπει να ενσωματωθούν και δεν μπορούν πια να γυρίσουν. Θα πρέπει λοιπόν εκεί που αναζητούν την προστασία να υπάρχει μια εργασία, να υπάρχει αυτή η πρόνοια. Νομίζω επίσης ε, ότι οι μειονότητες είναι ένα σημαντικό θέμα. Για μας δεν μου αρέσει και τόσο αυτή η λέξη βέβαια. Όμως νομίζω ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα μπορέσουμε επικοδομητικά να συνεργαστούμε και να τα πάμε καλά σε αυτό το επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα δίνω τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG Όχι, συγγνώμη. Πάμε στην ΚΟΕ. Σάντρα Περέιρα. Κυρία Περέιρα, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική έκθεσή της, κυρίως για το γεγονό ότι ανησυχεί ότι μειώνουν τα κονδύλια του Progress εκ μέρους του Συμβουλίου. Θέλουμε στα πλαίσια όλων των ταμείων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής Παγκοσμιοποίησης, των Ταμείων Υπέρ των Νέων, ε, και τα οποιοδήποτε ταμείο μπορεί να βοηθήσει τις ε, απόρους και να τους βοηθήσει να είναι ε, να έχουν πολλά κονδύλια δεδομένου ότι βοηθούν τους πιο ευάλωτες. Οι τροπολογίες τις οποίες εμείς καταθέσαμε πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα κονδύλια σε αυτά τα ταμεία. Κατά την άποψή μας, ο προπερισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να λάβει μέτρα τα οποία υποστηρίζουν τους εργαζόμενους με μέτρα, ε, τους προσφέρουν ε, εργασιακές σχέσεις σταθερές και προστούν να καταπολεμήσουν κοινωνικές ανισότητες. Το 2020 είναι το τελευταίο έτος του πενταετούς ε, πλαισίου Γι' αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και να μπορέσει στις γλωσσούς και να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Περέρα. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Στην κυρία Μπριζίτ Φελαχή, εκ μέρου τη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρο. Εκ μέρου τη Επιτροπή θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σα για τη γνωμοδότηση η οποία υποστηρίζει την πολιτική μας υπέρ της κοινωνικής ε, ε, ισότητας και της ε, απασχόλησης. Ξέρουμε ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει στα πλαίσια της πεντέτους πολιτικής μας το έτος επόμενο, που είναι το τελευταίο. Και βεβαίως έχουν γίνει πολλά υπέρ τη απασχόληση, αλλά δεν έχουμε κάνει αρκετά για να καταπολεμήσουμε την ένδια, τη φτώχεια. Επίσης, είπατε ότι πρέπει να εστιάσουμε προς την λήψη μέτρων που θα μπορέσουν να μας οδηγήσουν σε αποτελεσματικές πολιτικές. Θα ήθελα να πω ότι καταβάλουμε συνεχείς προσπάθειες, δεδομένου ότι είναι πιο δύσκολο να προσπαθήσει κανείς να εκτιμήσει τον αντίκτυπο πολιτικών και να δει ποια είναι τα αποτελέσματα και ελπίζουμε ότι στο πλαίσιο του προσεχούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου θα μπορέσουμε να είμαστε καλοί. Ξέρω ότι μας υποστηρίζετε στις προσπάθειες που καταβάλουμε. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση τώρα σε σχέση με αυτό το οποίο είπαν διάφοροι συνάδελφοί σας για το θέμα της ανεργίας των νέων. Ξέρουμε ότι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Ξέρουμε ότι οι προτάσεις της Επιτροπής αξιολογήθηκαν σωστά. Ξέρουμε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις ανάγκες κάθε κράτους μέλους και τη δυνατότητα απορρόφησης των κονδυλίων τα οποία δίδονται προς τους στόχους αυτούς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ να σε ενημερώσω λίγο για το χρονοδιάγραμμα. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών ε, είναι η 5η Σεπτεμβρίου το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 24 Σεπτεμβρίου. Σωστά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μπορούμε τώρα να περάσουμε στην ψηφοφορία. Καταρχάς, θα ψηφίσουμε με ανάταση της χειρός Ωστόσο όλοι σας θα πρέπει να έχετε την κάρτα ψηφοφορία σας. Μπορούμε να κάνουμε και μια επαλήθευση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με την τροπολογία 5650. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές ευχαριστώ τροπολογία 56-51 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται Περνάμε τώρα στροπολογία 56-52 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρτη ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Και η τροπολογία εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 56-53. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση και για αυτή την τροπολογία. Άρτη ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Και η τροπολογία εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 56-54. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 56-55. Εδώ θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. τροπολογία τώρα 56-57 καταπίπτει και περνάμε στην επόμενη 56-58 η οποία από ό,τι βλέπω έχει αποσυρθεί. Περνάμε έτσι στην τροπολογία 56-59. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται τροπολογια 5660 τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 56-61. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 56-62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 56-63. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5664. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 5665 καταπίπτει, δεν πρόκειται λοιπόν να την ψηφίσουμε. Και έτσι περνάμε στην 5666 υπέρ παρακαλώ. Α, σα δώσω συγγνώμη, λέει πρόεδρο. Καταπίπτει και η 5666. Ούτε και αυτή την ψηφίζουμε. Περνάμε στην τροπολογία 5667, λοιπόν. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Τροπολογία 5668, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 5669 56-69 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση, πολύ ωραία. Άρτη ψηφοφορία για την τροπολογία 5669. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Κύριε Πρόφη, όχι. Θέλετε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Πολύ ωραία, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, άρχεται εκ νέου ψηφοφορία Δεν είναι δυνατόν να το κάνουμε αυτό. Μάλιστα, με εξηγούν ότι δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τη ψηφοφορία και ούτε ήταν ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Περνάμε στην τροπολογία 5670, 5670 και 5671 από κοινού, παρακαλώ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 5672 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5673 Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5674. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5675. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την ε, τροπολογία 5675, άρτη ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Και η τροπολογία απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 5676, υπέρ παρακαλώ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5677, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. 5678 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 5686. Πρέπει να σας διαβάσω το διορθωτικό κείμενο το οποίο υπέβαλε η Γκουε, προφορική τροπολογία για την 5686, όπου λέγεται ότι το προτινόμενο σχέδιο θα εφαρμοστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην καλύπτει τις υφιστάμενες μελέτες που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή για την αξιολόγηση της ε, επερχόμενης πρωτοβουλίας όσον αφορά τους ελάχιστους μισθούς. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα, το πιλωτικό αυτό σχέδιο θα μπορούσε να προσφέρει μια προστιθέμενη αξία στις υφιστάμενες πρωτοβουλίες και θα μπορούσε να οδηγήσει, για παράδειγμα, σε μια πρωτοβουλία χαρτογράφησης των ε, ελάχιστων μισθών και αποδοχών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των προτάσεων που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 5684. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 5682 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονική επαλήθευση για την 5682 άρτη ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρασε Απορρίπτεται λοιπόν. Τροπολογία 56-90. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 56-93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία, μάλλον ηλεκτρονική επαλήθευση για την 5693 άρρηκτη ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5687 τώρα υπέρ κατά αποχές Μάλλον θα πρέπει να παληθεύσουμε το αποτέλεσμα ηλεκτρονικά, άρθρη ψηφοφορία και η τροπολογία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Και εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 5688. Νομίζω ότι έχουμε λάβει όλοι το διορθωτικό κείμενο μέσω προφορική τροπολογία. Είναι ιδιαίτερα εκτενέ το κείμενο, δεν θα το διαβάσω αυτή τη στιγμή. Γνωρίζετε το περιεχόμενο του κειμένου, έτσι δεν είναι. Πάλι πρώτε εδώ πέρα είναι να βελτιωθεί το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα βάσει των συστάσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5689 τώρα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 5681. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση και για αυτήν. Μάλιστα, λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία για την 5681. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5680 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5691 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονική επαλήθευση μάλλον και για αυτήν, άρτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 5685. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5679 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 56-94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Φτάσαμε έτσι στο τέλος των τροπολογιών. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, πολιτική απασχόλησης και κοινωνική πολιτική της ζώνης του ευρώ. Η κυρία Γιάννα Τόμ είναι η συντάκτρια της έκθεσης. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που θυμηθήκατε επίσης και πώς προφέρετε το επίθετό μου. Ευχαριστώ για την υποστήριξή τους γιατί δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο στη διαδεσία μας. Πρέπει να πω ότι οι συνθήκες στην ομάδα εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας προκαλούν αντιστοιχίες γιατί υπάρχουν ε, όσον αφορά το ποσοστό απασχόληση μεγάλες ε, ανισότητες, η ανεργία των νέων, οι συνθήκες εργασίας, η μακροχρόνια ανεργία, τα προβλήματα εξειδίκευσης, η έλλειπη προσόντων, η φτώχεια, η φτώχεια ακόμη και των εργαζομένων, οι συνήθικες εργασίες και όλα αυτά μας απασχολούν και δεδομένου ότι δεν έχουμε, είμαστε και σε καλή οικονομική κατάσταση, έχουμε ακόμη προβλήματα. Είδαμε τις συστάσεις και βλέπω ότι οι συστάσεις σε σχέση με το παρελθόν έχουν ε, ε κατά κάποιο τρόπο επιδεινωθεί. Ε, υπάρχει χαμηλό ποσοστό και ικανοποίησης και θα πρέπει να προσπαθήσουμε σε όλες τις χώρες να βελτιώσουμε τις συνθήκες, δεδομένου ότι η απασχόληση έχει σχέση και με άλλα οικονομικά μεγέθη και την υγεία των εργαζομένων. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε όλες αυτές τις τάσεις. Συγγνώμη κυρία Τόμ. Οι διερμηνείς Παρακαλώ να μην διαβάζετε με τέτοια ταχύτητα. Θα προσπαθήσω, λέει η συγγετρία. Και την ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκήσει πίεση στα κράτη-μέλη ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτέ τι στάσει. Διαφορετικά είναι άχρηστα όλα αυτά και οι μηχανισμοί που προβλέπονται. Οι ανισότητε στην ομάδα εργασία συνεχίζουν να υπάρχουν, όχι μόνο μεταξύ ε, ανδρών και γυναικών, αλλά διότι υπάρχει και αποκλεισμό των ατόμων που έχουν κάποια προβλήματα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει λοιπόν να βρουν λύσει στα προβλήματα αυτά. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν πολιτικές ε, συνειδητοποίησεις των προβλημάτων. Τα συστήματα κατάρτιση για όλους είναι απαραίτητα και έχουν αλλάξει οι συνθήκε σε όλες οι αγορέ εργασία πάρα πολύ. Παλιά κάποιος Είχε μια εργασία στην οποία ε, εξελισσόταν για διάρκεια τη επαγγελματική του καριέρα. Σήμερα αυτό ε, δεν υπάρχει. Πρέπει όλο και περισσότερο να εξειδικεύεται ο εργαζόμενο, να χρησιμοποιεί νέε μεθόδου, νέα εργαλεία, δεδομένου ότι η τεχνολογία τρέχει. Θα πρέπει όλοι λοιπόν να προετοιμαστούν ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ε, γρήγορα αυτέ τι αλλαγέ. Θα πρέπει να δούμε και πώς στα πλαίσια της εκπαίδευσης μπορούμε να κάνουμε κάτι. Οι διαφορετικά δεν θα μπορέσουν οι στόχοι, όσον αφορά τη μείωση του στόχοι, στα πλαίσια της πολιτικής για το 2020 να επιτευχθούν. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, τουλάχιστον 100 ε, εκατομμύρια πολίτες που ζουν σε κατάσταση ένδυας ή περίπου Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε και για αυτού. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να μας υποστηρίξουν στι τροπολογίε που καταθέσαμε οι συνάδελφοι. Ε, ελπίζω ότι στα πλαίσια της προθεσμίας που λύγει σύντομα θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο και συγγνώμη που μιλώ τόσο γρήγορα. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στους εισηγητές από μέρους του ΕΛΚ, η κυρία Walsh. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συνάδελφοι, χαιρετίζω την εργασία που έκανε η Συγγήτρια για την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητηθούν και οι κοινωνικές πτυχές απασχόλησης στην Ευρώπη. Πρέπει να κάνουμε και πολιτικές απασχόλησεις με ισχυρό κοινωνικό πρόθυμα. Θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των ανέργων αλλά κυρίως να εστιαστούμε στο θέματα που αφορούν την απασχόληση των νέων. Όσον αφορά τις κοινωνικές πολιτικές, υπάρχει ένας τομέας που με ενδιαφέρει όλο ενδιαφέρον και έχει εδώ παραγνωριθεί. Τα θέματα της ψυχικής υγείας των εργαζομένων. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλο αντίκτυπο και οικονομικό και κοινωνικό. Τα προβλήματα ψυχικής υγείας είναι πολύ σοβαρά και νομίζω ότι μπορούν να είναι καταστροφικά για τα άτομα τα οποία πάσχουν, για την οικογένειά τους, για τα άτομα που τα φροντίζουν και γενικότερα για την ε, κοινωνία. Πιστεύω ότι υπήρχαν και στο παρελθόν τέτοιου είδους προβλήματα όταν άρχισε η πεντετή του 2016 και ξέρουμε πόσο αντίκτυπο έχει σε όλους τους τομείς της ζωής τους και τις δυνατότητες που έχουν. Ξέρουμε ότι ε, πολλές φορές τα προβλήματα αυτά είναι τόσο σοβαρά και υποφέρουν τα άτομα τα οποία πάσχουν από κάποιο ψυχικό νόημα που στο τέλος οδηγούνται και σε αυτοκτονία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Το θέμα ψυχικής ε, υγείας είναι ένα γενικότερο πρόβλημα το οποίο επιδεινώνεται πολλές φορές από κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ώστε να προλάβουμε τέτοιου ισάρστα γεγονότα. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι και ελπίζω ότι στα πλαίσια του νέου προγράμματος θα, έχουμε, θα εστιαστούμε σε νέου είδους ενέργειες και δράσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα προγράμματα πρόληψης και συνειδητοποίησης ώστε να βοηθήσουμε τα άταρα τα οποία πάσχουν από τέτοιου είδους νοσήματα. Το κόστος επίσης πρέπει να πω ότι είναι σημαντικό για τα συστήματα υγείας και θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι διότι δεν υπάρχουν ε, επαρκή προγράμματα και πρωτοβουλίες στα πλαίσια αυτών των ατόμων. Σας ευχαριστώ και πάλι για την δουλειά που επιτελέσατε κυρία Εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. It's Mr. Nicholas Schmidt. Thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Γιάννα Τόμ, σωστά το είπα, για την έκθεσή της, αλλά και για τις ε, διευκρινήσεις που μόλις μας έδωσε. Νομίζω ότι ε, επιμένουμε πάρα πολύ στη θέση προτεραιοτήτων ε, επί των κοινωνικών θεμάτων και των θεμάτων απασχόλησης. Γιατί, Γιατί αν θέλουμε να έχουμε μια ευρωζώνη που είναι ισχυρή, θέλουμε και οικονομική και κοινωνική συνοχή και επίσης περιβαλλοντική συνοχή. Αυτό είναι και η αηφορία. Γι' αυτό πρέπει η έννοια της αηφορίας και της βιωσιμότητας να περάσει στη σκέψη μας και αυτό το έδειξε και το εξήγησε πολύ καλά και η πρόεδρος της Κομισιόν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο τελευταίο ευρωβαρόμετρο επίσης διαβάζουμε τις ανησυχίες των πολιτών. Όντως οι πολίτες θεωρούν ότι τα κοινωνικο-οικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα για αυτούς προσωπικά και θέλουμε μια Ευρώπη για όλους τους πολίτες, θέλουμε μια Ευρώπη που θα είναι στην υπηρεσία των πολιτών, ε, είναι τα πιο σημαντικά. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι πολλές ε, βελτιώσεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην απασχόληση, όμως παραμένουν ακόμα πολλά θέματα ανοιχτά. Οι ουλές της κρίσης δεν έχουν ακόμα υπουλωθεί, δεν έχουν ακόμα κλείσει. Είναι σημαντικό για την Επιτροπή μας λοιπόν να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα για την ευρωπαϊκή έρευνα ανάπτυξης έτσι ώστε να ενισχυθούν οι πολιτικές μας προς την κατεύθυνση μιας ανάπτυξης που περιλαμβάνει τους πάντες, να υπάρχει συνοχή και να υπάρχουν ποιοτικέ δουλειές με καλή αμοιβή για όλους. Επίσης, ευρέως συμφωνούμε με την αξιολόγηση του εισηγητή Θέλουμε όμως να τονίσουμε και τα μειονεκτήματα που ακόμη αντιμετωπίζουμε το ανέφερε και η κυρία Τόμ. Η μείωση της φτώχειας δεν ήταν τέτοια που θα περιμέναμε για το διάστημα μέχρι το 2020. Έχουμε συνεχώς αυξανόμενες ανισότητες στις κοινωνίες μας. Υπάρχουν μεγάλη, υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των κρατών μελών, αλλά όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών, α, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των περιφερειών και μάλιστα ως προς την ανεργία των νέων. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη, διότι είναι η δική μας αξιοπιστία έναντι των νέων που δοκιμάζεται. Πρέπει να μειώσουμε την ανεργία των νέων. Παραμένει μια πρόκληση. Αν δείτε τα ποσοστά, θα δείτε ότι σε λίγα κράτη-μέλη ε, δεν, είναι, δεν υπάρχει ε, ανεργία των νέων. Σε κάποια μάλιστα είναι πάνω από 30% ή και 40%. Επίσης αναφέρθηκε η έννοια της μετάβασης. Ε, ο κόσμος αλλάζει, όχι μόνο λόγω της τεχνολογίας, αλλά και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει λοιπόν να ενσωματώσουμε αυτή την ε, μετάβαση στις πολιτικές μας, στις οικονομικές, στις περιβαλλοντικές, στις φορολογικές πολιτικές μας. Όταν μιλάμε για μετάβαση πρέπει να τονίσουμε ότι η μετάβαση αυτή πρέπει να τους περιέχει όλους. Ναι, ταξιδέψουν μαζί μας όλοι οι πολίτες όλοι οι άνθρωποι. Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν πολλές ευκαιρίες, όμως ενέχουν και κάποιους κινδύνους. Μπορεί να είναι η πηγή επισφαλούς εργασίας, η κακής κοινωνικής προστασίας. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε συνοχή προς τα πάνω και όχι απλώς μετάβαση. Τώρα, η ανισότητα των φύλων. Υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις, αλλά ακόμα πόρο απέχουμε από τις κανονικές στοχεύσεις που είχαμε στην ατζέντα της Ρώμης. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τα εργαλεία μας ώστε να επιταχυνθεί η επίτευξη αυτών των στόχων. Ο κίνδυνος της ανέχειας αναφέρθηκε, χρειαζόμαστε νέα εργαλεία σε εθνικό επίπεδο που θα υποστηρίζονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να δούμε λίγο το ποσοστό τώρα της απασχόλησης. Όντως, παγκοσμίως υπάρχει βελτίωση. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί νέα προβλήματα να προκύψουν λόγω των οικονομικών δυσκολιών. Είναι σημαντικό λοιπόν και αυτό το θέμα. Θέλουμε επίσης να τονίσουμε τις πολιτικές ε, που ακολουθούνται για τους πιο ευάλωτους στην αγορά εργασίας. Το ανέφερε συνάδελφος ε, όχι μόνο οι μετανάστες, αλλά και τα άτομα με αναπηρία. Η απασχόληση των ατόμων με αναπηρία ε, είναι ακόμη ένα πρόβλημα. Η ενεργεία είναι υψηλή και δύσκολα μπορεί να βελτιωθεί το ζήτημα αυτό. Το, επίσης, στην διακήρυξη ΣΥΠΗ που πρόσφατα ε, είχαμε, οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων είπαν ότι πάντοτε θα υποστηρίζουν ε, την αρχή της δικαιοσύνης. Ε, είτε στην αγορά εργασίας, στην πρόνοια, στην οικονομία, στην ψηφιακή μετάβαση, είτε πρόκειται ε, για το ένα είτε για το άλλο θέμα, ε, αυτή είναι η δέσμευσή τους. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε πολύ για να μειώσουμε τα κενά που υπάρχουν. Ευχαριστούμε πολύ για τους πράσινους. Κύρα Πέτερ Χάνσεν. Ναι, ευχαριστώ να σας ευχαριστήσω για το ε, σχέδιο της έκθεσης ε, να τονίσω ότι για τους πράσινους οι κοινωνικές δεσμεύσεις και στόχοι είναι το ίδιο σημαντικοί με τους οικονομικούς. Πρέπει πραγματικά να έχουμε μια μεταμόρφωση της κοινωνικής διάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε ένα δίκαιο και σταθερό ε, περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι πρέπει να επενδύσουμε στην απανθρακοποίηση, ιδιαίτερα στην βιομηχανία και στον ενεργειακό τομέα. Επίσης, θα μιλήσω για τους αυτοαπασχολούμενους και τους μη μισθωτούς, ε, όπως και για τους άστεγους. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αδειμονώ για μια ε, επικοδομητική συνεργασία με όλους σας. Ήσασταν γρήγοροι, ευχαριστούμε για τη δημοκρατία και την ταυτότητα. Υπάρχει κάποιος. Όχι, δεν έχω κάποιο όνομα εδώ, ούτως ή άλλως. Ωραία, για το ECR, η κυρία Ραφάλσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση αυτή, να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για τις σαφέστατες αυτές τις πληροφορίες που μας έδωσε, που αγγίζουν πραγματικά τα πιο κέρια προβλήματα όσον αφορά την πολιτική απασχόληση. Μία σωστή όμως πολιτική απασχόληση, σας μην το ξεχνάμε, είναι καθοριστική σημασία προκειμένου όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί προς τον σωστό δρόμο. Σαφώς, πολλά προβλήματα αντιμετωπίζουμε στο τομέα της απασχόλησης, προβλήματα τα οποία τόνισαν και οι προλαλήσαντες. Ωστόσο υπάρχει μια πτυχή την οποία δεν φωτίσαμε αρκετά. Ποιότητα της εργασίας, η ηθική, η ιδεοντολογία στα πλαίσια της απασχόλησης και της εργασίας, η ασφάλεια και η προστασία, αλλά ακόμα και το κόστος της εργασίας. Νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την απασχόληση σε όλες αυτές τις πτυχές χωρίς να δαπανίσουμε πάρα πολλά κονδύλια. Α μην ξεχνάμε επίση ότι τίθεται το ζήτημα τη μη διακριτική μεταχείρισης στο πλαίσιο τη απασχόληση. Και για το ζήτημα αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αποδοτικά και αποτελεσματικά εργαλεία, μεθόδου και μέσα ουσιαστικά που έχουν οδηγήσει σε επιτυχία στο παρελθόν. Α μην ξεχνάμε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια μιλάμε για την εγγύηση για του νέου, για την απασχόληση των νέων. Εκεί όμω δεν είδαμε τα αποτελέσματα και μπορούμε να μιλήσουμε ακόμα και για φιάσκο βλέπουμε ότι η ανεργία, ιδίω ανάμεσα στους νέους, μπορεί να παρουσιάζει μια μηδαμινή μείωση για κάποιες χώρες, αλλά παρόλα αυτά παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Η αγορά εργασίας εν γέννη στην Ευρώπη λέγεται ότι βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Ε, α, εποφεληθούμε λοιπόν από την θετική αυτή συγκυρία, εποφεληθούμε από από τα νέα μέσα Ενημέρωση, επικοινωνίε, καθώ επίση και από τι νέε τεχνολογίε προκειμένου να βελτιώσουμε τα επίπεδα απασχόληση. Α μην ξεχνάμε όμω ότι η ίδια η φύση της εργασίας θα τροποποιηθεί, θα μετασχηματιστεί στο μέλλον. Α είμαστε λοιπόν και εμεί έτοιμοι για τι σημαντικέ αυτέ αλλαγέ. Βλέπουμε ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη κινητικότητα στο τομέα τη απασχόληση, ότι θα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερε καινοτόμε τεχνολογίε αλλά μην ξεχνάμε ότι οι τεχνολογίες αυτές θα αλλάξουν άρδιν την ίδια τη φύση της απασχόλησης. Επίσης, θεωρώ ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την όλη ευελιξία που προτείνεται τώρα για τον τομέα της εργασίας. Θα πρέπει όμως και αυτή να χρησιμοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουμε τελικά μια απασχόληση η οποία θα είναι σωστή. Η κυρία Περέρα έχει το λόγο του της ΓΚΟΕ, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο για την έκθεσή της. Και εμείς ε, μπορούμε να συμμεριστούμε τις ανησυχίες της για την ανεργία των νέων, για την ε, φτώχεια των εργαζομένων, για την ε, ανάγκη να κάνουμε θέσεις εργασίας καλής ποιότητας και να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων και όλες τις άλλες. Θα πρέπει στα πλαίσια της ε, ευρωπαϊκής οικονομικής διαχείρισης να γίνει μια προσπάθεια ώστε να καταπολεμηθούν αυτά τα φαινόμενα. Οι πολιτικές ε, απασχόλησης και οι κοινωνικές πολιτικές, έτσι όπως τις έχει ψηφίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουν ε, οδηγήσει σε βελτίωση της αγοράς εργασίας, αλλά σε αποσταθεροποίηση έχει οδηγήσει στο να παγώσουν οι αμοιβέ και έχει δημιουργήσει κοινωνικά προβλήματα και ανισότητε μεταξύ των εργαζομένων. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι ώστε να μπορέσει η κοινωνική πτυχή του προβλήματος να ενισχυθεί, να μπορέσουν οι ειδικέ συστάσεις να εφαρμοστούν από όλους για να μην μιλούμε για τις ε, ανισότητες που υπάρχουν στα πλαίσια των πολιτικών που εφαρμόζονται και μειώνουν όλο και περισσότερο τα κοινωνικά ε, ε, την οποιαδήποτε κοινωνική πολιτική. Στην Πορτογαλία δεν εξεχάσαμε την ε, άσχημο θέαμα το οποίο δημιουργήθηκε και τις απειλές που ε, δημιουργήθηκαν ώστε να αφήσουμε κατά μέρος τις ε, πολιτικές μας και να ακολουθήσουμε πάντα τις πολιτικές που επέβαλε η Τρόικα. Μπορέσαμε να κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει όλες οι πολιτικές να εφαρμόζονται πάντα με κοινωνικό πρόσημα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπλεγκαβιτσιούτε ζήτησε το λόγο. Ναι, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, διότι στην έκθεσή της συμπεριλαμβάνονται πάρα πολλά προβλήματα, πράγμα που αποδεικνύει πόσο σημαντικές είναι οι διάφορες πτυχές της ε, πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας στα προβλήματα για τα οποία ήδη έχει αρχίσει να εργάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε ότι θα ασχοληθεί πολύ σοβαρά με αυτά τα προβλήματα η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των εργαζομένων όλων όσον αφορά διάφορες ανισότητες μεταξύ των αμοιβών ανδρών και γυναικών μεταξύ άλλων προβλημάτων που δεν μπορέσαμε να βελτιώσουμε με λύσεις σωστές. Θα πρέπει λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνει κάτι ώστε να βελτιωθούν τα πράγματα. Δεύτερον, η απασχόληση των νέων, η ανεργία που πλήττει τους νέους. Έχουμε ένα αποτελεσματικό μέσον που είναι η εγγύηση για την ε, νέους μπορούμε με διάφορες πολιτικές να βελτιώσουμε τις συνθήκες απασχόλησης των νέων. Αλλά πρέπει να πω ότι το επίπεδο ανεργίας σε κάποια κράτη-μέλη είναι πολύ υψηλότερο από το μέσο ευρωπαϊκό ε, επίπεδο. Άρα οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούμε δεν είναι πάντα αποτελεσματικοί. Η φτώχεια, η ένδυα επίση είναι σοβαρό το πρόβλημα. Η φτώχεια των εργαζομένων που εργάζονται όμως με κακές συνθήκες και κακή αμοιβή. Είναι γενικότερο πρόβλημα. Σχοληθήκαμε εδώ και χρόνια με το θέμα αυτό, αλλά δεν μπορέσαμε να βελτιώσουμε την αμοιβή των νέων. Δεν τους δίνουμε και κοινωνικά βοηθήματα αρκετά ώστε να μπορέσουν να ζουν με αξιοπρέπεια. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια κατώτατη αμοιβή ώστε να ζουν αξιοπρεπώς οι άνθρωποι. Έχουμε πάρα πολλά έγγραφα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στα οποία λέμε ότι θα μπορέσουμε την ανεργία των νέων να την εκριζώσουμε. Τα παιδιά, πολλά παιδιά ζουν σε κατάσταση ένδυα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό, ότι εκτός από τα εθνικά προγράμματα θα πρέπει να θεσπίσουμε και να εφαρμόσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα, κυρίως για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά της ε, θα ήθελα να πω το εξή στην εκπρόσωπο τη Επιτροπή. Κάνει συστάση η Επιτροπή που υποβάλλει στα κράτη-μέλη όσον αφορά την κοινωνική πολιτική το τι μπορεί να βελτιωθεί, την πολιτική απασχόληση, αλλά εν τρίτο των χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να θέσει σε εφαρμογή αυτέ τι συστάσει. Για ποιο λόγο λοιπόν τι εκπονεί τι συστάσει η Επιτροπή, αν κανένα δεν τι εφαρμόζει. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε τα κράτη-μέλη να, σε, να κάνουν πράξη αυτές τις συστάσεις. Διαφορετικά δεν κάνουμε τίποτε. Πέντε χρόνια θα περάσουν ακόμη και θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών μας. Θα ήθελα και πάλι να συγχαρώ την εισηγήτρια, τους σκιώδεις εισηγητές και ελπίζω ότι η εργασία που θα επιτελέσουμε από κοινού τα επόμενα πέντε χρόνια θα καταλήξει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και θα έχουμε νομοθετικά κείμενα που θα μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε την κατάσταση όλων των πολιτών της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Νικόλας Αλαβάνο. Ευχαριστώ, ε, κυρία Πρόεδρε. Σε σχέση με την έκθεση με την οποία ανταλλάσσουμε απόψεις, είναι ζήτημα να εξεταστούν ε, οι όροι εργασία στο σύνολο των εργαζομένων για να βγει συμπέρασμα, καθώ η στατιστική με την οποία δουλεύει η έκθεση ανακατεύει του μόνιμου εργαζόμενου με τη μερική απασχόληση, ακόμη και εκείνους που κάνουν δύο-τρία μεροκάματα το μήνα και του βαφτείς γενικά απασχολούμενου. Σχετικά με τον αριθμό των απασχολούμενων συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχέση μεταξύ σταθερή και μερική απασχόληση, στοιχεία τα οποία δίνουν οι διεθνείς οργανισμοί για το 2018 δείχνουν αντίθετη πορεία. Ότι αυξάνεται η μερική απασχόληση και έχει ξεπεράσει συνολικά το 1 τρίτο των απασχολούμενων. Η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε σε μία σειρά από χώρε δείχνει ότι οι αποδοχές για το μέσο μισθό απολύτως μειώνονται σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και της λογικής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που συμπιέζουν το σύνολο των δικαιωμάτων των εργαζομένων προς τα κάτω. Αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης, ξεπερνώντας τα 67 έτη στη λογική της ενεργού γύρανσης και της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών ταμείων, πράγμα το οποίο και η παρούσα έκθεση το διαπιστώνει όταν δείχνει ότι αυξάνεται η απασχόληση για τους ανθρώπους άνω των 55 ετών. Αντίστοιχα, διαπιστώνει η έκθεση το σοβαρό πρόβλημα τη νεανική ανεργία, αλλά ποια είναι η λύση που προτείνει. Κινητικότητα και επιχειρηματικότητα των νέων. Δηλαδή, η λύση είναι τα εκατομμύρια των νέων ανέργων τη Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνουν επιχειρηματίε. Η πανάκια η οποία προτείνει η έκθεση στην πραγματικότητα είναι η αυστηρότερη εφαρμογή των εξειδικευμένων συστάσεων κατά χώρα τη Κομισιόν. Μέτρα δηλαδή που όχι μόνο δεν θωρακίζουν και διευρύνουν την πλήρη απασχόληση με αξιοπρεπή μισθό και δικαιώματα, αλλά αντίθετα, όπω ήταν και στην κατάσταση που, ε, που έχουμε στη χώρα μας, στην Ελλάδα, γενικεύουν την ελαστική απασχόληση. Κόβουν δικαιώματα στη λογική της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της μείωσης του εργασιακού κόστους. Αφοπλίζουν τους εργαζομένους, κάνοντας δυσκολότερες τις διεκδικήσεις τους. Νομοθετούν ενάντια στην απεργία, απελευθερώνοντας τις απολύσεις, κάνοντάς τες και ευκολότερες με πρόσχημα τα προσωπικά δεδομένα. Κατά την άποψή μας πρόκειται για έκθεση που έχει στόχο να ωρεοποιήσει από τη μία την άσχημη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι μέσα στου τόπου δουλειά, αλλά και την ίδια την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που για να θωρακίσει τα συμφέροντα των μεγάλων ομήλων, ρίχνει στην άβυσο μισθού, συντάξει, δικαιώματα. Και εκφράζουμε την έντονη διαφωνία μα. Η λύση είναι οι εργαζόμενοι, οι απασχολούμενοι σε όλου του κλάδου, με οργανωμένο τρόπο μέσα από τα συνδικάτα του, με ταξικό προσανατολισμό, να βάλουν πλώρη για αιτήματα, δικαιώματα και μισθού στο ύψο των σημερινών σύγχρονων αναγκών τους. Ευχαριστώ πολύ. Now, Gualmini. Η κυρία Γουαλμίνη τώρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω καταρχάς την εισηγήτρια, την κυρία Γιάννα Τόμ, διότι νομίζω ότι ε, το σχέδιο ψηφίσματος προτείνει είναι πολύ θετικό και ιδιαίτερα ευρύ. Καλύπτονται δηλαδή πολλά ζητήματα προβληματικά που έχουν να κάνουν με την ε, αγορά εργασίας. Επομένω θεωρώ ότι αυτό από μόνο το αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα, προκειμένου να καταφέρουμε να ενισχύσουμε τη δράση της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα συγκεκριμένα αυτά προβληματικά ζητήματα. Τώρα πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να τονίσω μία συγκεκριμένη πτυχή που νομίζω ότι αποσιάζει από την πρόταση ψηφίσματος της εισηγήτριας και μάλιστα ως προς αυτό θα ήθελα να καταθέσω και μια σειρά από τροπολογίες. Ξέρω ότι η προθεσμία είναι η 5η Σεπτεμβρίου, πάντως σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο λείπει από την έκθεση αυτή και είναι αυτό που έχει να κάνει με τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, τα δημόσια γραφεία απασχόλησης. Όπως γνωρίζετε, τα αποτελέσματα στον τομέα της απασχόλησης τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον τονίζουν όλο και περισσότερο ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τον συνεχή εξυγχρονισμό αυτών των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης και μάλιστα να καταφέρουμε τρόπον την να εναρμονίσουμε και τις δημόσιες αυτές υπηρεσίες απασχόλησης έβρεση εργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να προσφέρουμε την κατάλληλη κατάρτιση στους δημόσιους υπαλλήλους που απασχολούνται στις υπηρεσίες αυτές προκειμένου πραγματικά να μπορούν να ταποκριθούν στις προκλήσεις και τα προβλήματα της ε, υφιστάμενης ε, αγοράς απασχόλησης. Θα υποβάλω λοιπόν κάποιες σχετικές τροπολογίες ελπίζω ότι θα γίνουν δεκτές και από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες. Θεωρώ ότι οι οροπολικές αυτές έχουν ένα οριζόντιο χαρακτήρα. Τονίζω ότι χρειαζόμαστε δημόσιες τέτοιες υπηρεσίες, οι οποίες να μην λειτουργούν μόνο για τις μειονεκτούσες κατηγορίες αγοράς εργασίας, αλλά χρειαζόμαστε αποτελεσματικές και μοντέρνες τέτοιες υπηρεσίες απασχόλησης για κάθε επαγγελματική κατηγορία και για κάθε δαφικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Κυρία Μπέσοφ τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήδη γίνανε πολλές παρατηρήσεις ε, για την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι ε, η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για την Επιτροπή μας. Είμαστε πάρα πολύ καλοί στην ανάλυση που κάνουμε εν γέννη, αλλά αυτό που μας λείπει θα έλεγα συνήθως είναι να καταλήγουμε σε κάποιες πιο σαφείς και συγκεκριμένες συστάσεις. Νομίζω λοιπόν θα μπορούσαμε εδώ πέρα να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση. Συμφωνώ με την πρόταση που γίνεται ότι οι επενδύσει είναι κέρια σημασία και νομίζω ότι θα έπρεπε εδώ πέρα να επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο στι επενδύσει κοινωνική φύση. Και κάτι που λείπει επίση από την έκθεση είναι το εξή. Πολύ ωραία, μιλάμε για ποιοτική και αξιοπρεπή εργασία, αλλά θα πρέπει να καταφέρουμε να ενισχύσουμε και τις λογικές συμβάσεις και ως προς αυτό χρειαζόμαστε και μέτρα ενωσιακά, από το κοινωνικό δηλαδή επίπεδο. Νομίζω ότι αν προσθέσουμε και τα στοιχεία αυτά, η έκθεση θα γίνει πολύ καλύτερη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Προτού προχωρήσουμε, θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις με την άδειά σας βέβαια. Άκουσα προσεκτικά τα όσα είπαν οι προαλήσαντες και κάτι το οποίο λείπει από τη συζήτηση αυτή κατά την άποψή μου είναι ένα βασικό πρόβλημα. Γνωρίζουμε ποια είναι τα βαθύτερα αίτια της πολύ υψηλή ανεργίας των νέων, γιατί προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα, να έχουμε δηλαδή μειωμένη ανεργία για τους νέους, να καταφέρουμε να μειώσουμε τους τεράστιους αυτούς αριθμού, τα τεράστια αυτά ποσοστά ανεργίας των νέων, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να λύσουμε ποτέ το πρόβλημα αν δεν γνωρίζουμε τα βαθύτερα αίτια. Για ποιο λόγο δεν απασχολούνται περισσότερο οι νέοι από του εργοδότε, αυτό που μου λένε οι εργοδότες συνήθως είναι ότι φταίει το εκπαιδευτικό σύστημα, ότι πολύ συχνά οι νέοι δεν είναι έτοιμοι να αναλάβουν μια εργασία, ότι δεν είναι έτοιμοι να αναλάβουν επαγγελματικά καθήκοντα και γι' αυτό το λόγο οι εργοδότες λένε ότι δεν είναι έτοιμοι να τους απασχολήσουν. Αν θέλουμε λοιπόν να λύσουμε το ζήτημα αυτό, ενδεχομένως δεν θα πρέπει να πιέζουμε μόνο για καλύτερη χρηματοδότηση από τα κοινοτικά ταμεία, για πιο αποτελεσματική χρήση των ταμείων αυτών, Ίσως θα έπρεπε να ενσωματώσουμε και κάποιες ε, προτάσεις που να έχουν να κάνουν με την ίδια την εκπαίδευση και την κατάρτιση των νέων. Για παράδειγμα, καλύτερη επαγγελματική καθοδήγηση για τους νέους, ε, καλύτερη κατάρτιση των διδασκόντων, των υπεύθυνων για την εκπαίδευση δηλαδή των νέων, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι θα είναι πιο έτοιμοι να αναλάβουν μια επαγγελματική θέση, θα είναι πιο έτοιμοι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Αυτή ήταν η σύντομη παρατήρηση που είχα να κάνω εγώ όσον αφορά τώρα το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 5η Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Σας παρακαλώ να καταθέσετε τροπολογίες μόνο στην αγγλική γλώσσα και μόνο μέσω email. Στις 2 και 3 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας εν συνεχεία. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Γιούτε, από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λίγα ε, σχόλια για την έκθεση. Ε, πριν ξεκινήσει ε, η νέα Επιτροπή τη θητεία της. Καταρχάς, να σκεφτούμε λίγο την κατάσταση στους τομείς της απασχόλησης ε, και των κοινωνικών πολιτικών. Έχουν πολλά επιτευχθεί, απασχόληση, μείωση της φτώχειας, ε, όμως ε, πολλά πράγματα παραμένουν μη ακανοποιητικά όπως όλοι γνωρίζουμε, παρά την πρόοδο. Η έκθεση επίσης δείχνει πώς ε, η Επιτροπή Γιούγκερ προσέγγισε τις πολιτικές, όπως τον Ευρωπαϊκό Σπυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ο στόχος ήταν η συνοχή για τις ε, ε, συγκεκριμένες συστάσεις αναχώρα. Η Επιτροπή συμμερίζεται τα ποσοστά εφαρμογής, όμως τονίζεται ότι η εφαρμογή μέτρων που επηρεάζουν την ζωή των ανθρώπων χρειάζεται χρόνο δεν είναι μόνο τα κοινοβούλια και οι θύνοντες που αποφασίζουν. Πρέπει να εφαρμοστούν σε ανθρώπους αυτά και αυτό συχνά το ξεχνάμε. Γενικά το σύστημα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και οι συγκεκριμένες συστάσεις σε χώρα έχουν ουσιαστική επίπτωση στην διαμόρφωση πολιτικών και τις μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη. Για να καταλήξω να πω ότι πολλά στοιχεία της έκθεσης ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές οδηγίες και τις κατευθυντήρες γραμμές που έδωσε η κυρία Φοντερ και αυτά που είπε και ο κύριος Σμιτ. Ελπίζω ότι στα επόμενα χρόνια θα συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό. Τώρα, η κυρία Τόμ, έχετε τον τελικό λόγο. Ευχαριστώ, συνάδελφοι, για αυτή τη συζήτηση. Κάποιες φορές αν ε, ε, εγκρίνεις ε, κάτι, μόνο οι σκιώδεις μιλούν, αλλά όταν μιλάνε και άλλοι είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ λοιπόν. Είχαμε ένα όριο 6.000 χαρακτήρες για τις τροπολογίες. Θα κάνω μόνη μου κάποιες, ένα κλέψιμο ας πούμε κάνω. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας και για την πολύ καλή συζήτηση. Thank you. Now we will continue with the... Να συνεχίσουμε με την ανταλλαγή απόψεων τώρα με τον Γιώργο Κόρτε, που είναι ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης ΕΜΠΛ. Τον καλωσορίζουμε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Κόρτε, μπορείτε να μας κάνετε την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε εδώ σήμερα τώρα ε, που ξεκινάτε τις συναντήσεις της Επιτροπής σας. Είναι μεγάλο προνόμιο για μένα που έρχομαι εδώ για να σας παρουσιάσω τις βασικές δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσής μου και να σας ενημερώσω για τους βασικούς ε, τομείς πολιτικής για τους οποίους είμαστε υπεύθυνοι ε, στο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ξεκινήσω λέγοντας πόσο σημαντική υπήρξε αυτή η Επιτροπή τα τελευταία πέντε χρόνια. Ε, πέρασε μια πολύ φιλόδοξη ατζέντα που εφάρμοσε ο πρόεδρος ε, Γιούγκερ και η Μαριάννα Τάισεν, η, Επιτροπή, η Επιτροπός μας. Και από την εμπειρία μου τους τελευταίους 18 μήνες να σας πω ότι δεν θα ήταν εύκολο ε, για μας να εγκρίνουμε και να εφαρμόσουμε τόσο σημαντικά θέματα χωρίς τη δική σας ε, βοήθεια. Χρειαζόμαστε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα έχω πάντοτε καλή ανάμνηση όλων αυτών των έντονων στιγμών που περάσαμε στις τριμερείς ε, διαπραγματεύσεις ε, και στις συζητήσεις μας. Δεν έχω σκοπό τώρα, σήμερα το πρωί, να σας κάνω ένα ταξίδι στην κάθε μία ξεχωριστή δραστηριότητά μας θα ήταν ιδιαίτερα βαρετό και θα χρειαζόμασταν και ώρες. Δεν είναι χρήσιμο. Η Γενική Διεύθυνση ε, έχει ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Ε, γι' αυτό ζήτησα από τους διευθυντές μας να έρθουν εδώ. Ε, είναι εδώ στην αίθουσα σήμερα και θα είναι στη διάθεσή σας για πιο άμεση επικοινωνία με σας ή τους και τις βοηθούς σας να επικεντρωθώ λοιπόν εγώ στις ε, κέρυες δραστηριότητές μας, στις βασικές δραστηριότητές μας και να αφήσω μετά χρόνο σε εσά για ερωτήσεις. Καταρχάς θα πω μερικά λόγια για τη Γενική Διεύθυνση, ε, της οποίας είμαι Γενικός Διευθυντής και μετά θα σας πάω ε, στα τέσσερα μπλοκ ε, της ε, δραστηριότητάς μας. Πρώτον, η νομοθεσία. Δεύτερον, ευρωπαϊκό εξάμεινο. Τρίτον, τα κονδύλια. Είμαστε υπεύθυνοι για το 10% του δημοσιονομικού πλαισίου, πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Επίσης, έχουμε τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία. Σε αυτά θα επικεντρωθώ να δώσω όμως μια σύνοψη ε, των δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και θα το κάνω στα γαλλικά. Έτσι λοιπόν, επιτρέψτε μου καταρχάς ε, να περάσω στα γαλλικά και σύντομα να σας παρουσιάσω τη γενική μου διεύθυνση. Η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης ε, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή Όλα αυτά για την πρόθεση της ελεύθερης διακίνησης των πολιτών και την πρόθεση των κοινωνικών ε, μέτρων και να μπορέσουμε να κάνουμε μια σωστή κοινωνία. Οι στόχοι μας λοιπόν είναι αρκετά φιλόδοξοι. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι είμαστε υπό την ε, υποπτία της Επιτρόπου Μαριαν Τάισεν και με ευχαριστήσει Συνεργαζόμαστε και με τον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκης και βεβαίως εργαζόμαστε και απευθείας και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η πολιτική τους, οι προσανατολισμοί τους και ο ενθουσιασμός τους επέτρεψαν η κοινωνική πολιτική πολιτική απασχόλησης να είναι σε ένα το υψηλότερο επίπεδο. Η γενική μας διεύθυνση πρέπει να σας πω ότι απασχολεί περίπου 900 άτομα σε 7 διευθύνσεις και 37 μονάδες. 37, ε, από τις 37, 36 βρίσκονται στις Βρυξέλλες σε τρία διαφορετικά κτίρια και μόνο μία βρίσκεται στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για την ομάδα ασφάλεια στην εργασία και υγεία. Έχουμε κυκλοφορήσει ένα δελτίο με τις ε, κύριες πληροφορίες που αφορούν τα καθήκοντά μας ως γενική διεύθυνση. Και Κυρίως μιλώ για, κύρια, για πέντε ουσιαστικά καθίσματα που έχουμε. Ε, είμαστε υπεύθυνοι για την κοινωνική ανάλυση, για την νομοθεσία, για τις αρμοδιότητες, skills, για την επαγγελματική κατάρτιση, για την διαχείριση των ταμείων και των κονδυλίων που χειριζόμαστε και για την απαλλαγή από τους υπεύθυνου ε, στα θέματα οικονομικά, εσάς και το ελεγκτικό συνέδριο. Πρέπει να σας πω ότι διαχειριζόμαστε περίπου 13,5 δις ευρώ ετησίως. Έχω ε, νέα country desk σε, ε, τα πλαίσια των 28 κρατών μελών και έχουμε και μία ε, διεύθυνση Οικονομικού Ελέγχου. Για να χειριστούμε λοιπόν σωστά αυτά τα 13,5 δις. 10 λοιπόν το 100 περίπου του κοινοτικού προϋπολογισμού. Και τελικά η Γενική μας Διεύθυνση είναι υπεύθυνη και για 5 ευρωπαϊκούς αποκεντρωμένους οργανισμούς. Θα σας πω τα ονόματά τους αγγλικά διότι έτσι τους ε, γνωρίζουμε όλοι. Στα αγγλικά λοιπόν. Πρώτος οργανισμός, το Eurofound, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τις Συνθήκες Εργασίας και Διαβίωσης στο Φλωρίδα, η όσα στο Μπιλμπάο για την ασφάλεια στην εργασία, το ΣΕΝΤΕΦΟΠ στη Θεσσαλονίκη, στο Τουρίνο το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κατάρτισης, και το πιο πρόσφατο την ε, αρχή για θέματα εργασίας που θα έχει ως έδρα την Πρατισλάβα. Ποιε είναι οι κυρίες δραστηριότητες λοιπόν. Τι απασχολεί αυτά τα 900 άτομα στην καθημερινότητά τους. Όπως σας είπα θα είναι χρήσιμο για σας να το ε, σας παρουσιάσω τέσσερις κύριους τομείς. Την νομοθεσία, το ευρωπαϊκό εξάμεινο, τα κοινοτικά ταμεία και το κοινωνικό διάλογο. Πρέπει να σας πω τώρα ότι τα τρία θεσμικά όργανα το 2017 στο Λουξεμβούργο υποστήριξαν τον πυλώνα το, βάσει του οποίου εμεί εργαζόμαστε στα πλαίσια των κοινωνικών δικαιωμάτων, στα πλαίσια της κοινωνικού χάρτη και νομίζω ότι έχετε στη διάθεσή σας αντίγραφο του ε, τι, ακριβώς του εγγράφου που ασχολείται με τα θέματα αυτά στα πλαίσια του πυλώνα μας απασχολεί για τα κοινωνικά θέματα και νομίζω ότι είναι χρήσιμο να το εγγράψετε. Τι κάνει λοιπόν ο πυλώνας. Εκφράζει συλλογικά 20 αρχές που πρέπει να εφαρμοστούν για να μπορούν να λειτουργούν σωστά οι τομείς απασχόλησης κοινωνικής πολιτικής. Αυτός ο πυλώνας σε πράξη δεν είναι μόνο θέμα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά όλων των κρατών, μελών, των κοινωνικών εταίρων και των υπολείπων ευρωπαϊκών ε, ε, οργάνων. Και η νέα πρόεδρος της Επιτροπής έχει αναλάβει δεσμεύσεις για την πλήρη εφαρμογή του. Και πρέπει να σας πω ότι όχι μόνον η πρόεδρος της Επιτροπής έχει αναλάβει τέτοιες δεσμεύσεις, αλλά και όλοι οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων και εκπρόσωπος του Συμβουλίου έχουν αναλάβει δεσμεύσεις, ώστε στα πλαίσια της νέας στρατηγικής ατζέντας που εγκρίθηκε τον Ιούνιο, τον Ιούνιο φέτος, να εφαρμόσουν τις αρχές αυτές. Βεβαίως δεν δόθηκε μεγάλη δημοσιμιότητα στο γεγονός, δεδομένου ότι υπήρχαν άλλα πολιτικά γεγονότα, αλλά πρόκειται για ε, μία δέσμευση πολύ σημαντική εκ μέρου των κρατών μελών. Τι κάνει λοιπόν αυτός ο πυλώνας. Εμπνέει όλους αυτούς οι οποίοι πρέπει να εφαρμόσουν αυτές τις πολιτικές. Πρώτα απ' όλα, στον τομέα που μας απασχολεί, πρώτα απ' όλα η νομοθεσία. Είναι σημαντικό να σας εξηγήσω εν συντομία ότι υπάρχουν διάφορες ε, ε, διατάξεις στα πλαίσια της ε, Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση νομοθεσίας. Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και καλύπτουν όλους τους τομείς. Πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για ένα σύνολο κανόνων πολύ πολύπλοκων. Αλλά η συνθήκη είναι αυτή η οποία θεσπίζει κάτι τέτοιο. Βεβαίω, όταν πρόκειται για την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων, το άρθρο 45 είναι σαφές τι λέγεται στα πλαίσια τη ενιαία εσωτερική αγοράς και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίζει την άρση οποιοδήποτε ε, εμποδίου για την μετακίνηση των εργαζομένων. Το 48 επίση είναι άρθρο, είναι πολύ σημαντικό. Νομική βάση για το συντονισμό των, ε, συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης κρατών μελών. Αυτό είναι το θέμα το οποίο θα σας αναφέρει στις 5 η κυρία Τάισεν. Πρόκειται για τη νομική βάση που αφορά τον ε, κανονισμό που διέπει το θέμα αυτό. Είναι σημαντικό να πούμε ότι πρόκειται για συντονισμό της νομοθεσίας που αφορά τα κοινωνικά συστήματα και όχι για ε, εξίσωση όλων των συστημάτων. Συντονισμό. Και αυτό είναι κάτι είπα, που θα το συζητήσετε σήμερα το απόγευμα. Το άρθρο 45, το 48 είναι διατάξεις πάρα πολύ σημαντικές. Υπάρχει και το 153 για τις κοινωνικές πολιτικές που είναι επίσης σημαντικό και σας συνιστώ να το μελετήσετε. Πρόκειται για μια σημαντική ε, διά, διάταξη που λέγει ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίζει σε κάποιου τομεί τι πολιτικέ τι οποίε θέτουν σε εφαρμογή τα κράτη-μέλη. Και στα πλαίσια τη πολιτική το 153, 54 και 55 είναι πολύ σημαντικά και θα μπορούσα να σας κάνω ολόκληρο σεμινάριο για να σας τα εξηγήσω, γιατί πρόκειται για νέες διατάξεις πολύπλοκες. Συνοπτικά, τι λέει, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ένωση μπορεί να θεσπίσει κατώτατα όρια τα οποία θα πρέπει να σέβονται όλα τα κράτη-μέλη σε όλες τις πολιτικές. Σύνθηκες εργασίες κοινωνικά συστήματα, κοινωνική προστασία των εργαζομένων, θέματα υγείας και προστασίας των εργαζομένων, ε, ενημέρωση, διαβούλευση και ε, συνθήκες για να περιληφθούν στην αγορά εργασίας όσοι αποκλείονται, για να μην αποκλείεται κανείς. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για να μπορέσει κανείς να προχωρήσει περισσότερο και είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια των συζητήσεων που γίνονται για να κατανοήσουν όλοι περί τίνος πρόκληση, διότι πρόκειται, διότι υπάρχουν πάρα πολλές παρανοήσεις σε επίπεδο κρατών μελών. Θέτουμε λοιπόν εμείς τα θεμέλια, το κατώτατο όριο, κάτω από το οποίο δεν μπορεί κανείς να κατέβει. Επίσης, στα πλαίσια των κοινωνικών πολιτικών υπάρχουν και άλλα θέματα. Όταν όμως νομοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακολουθεί πολιτική ανάλυση βάση αποδείξεων και μαρτυριών, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη νομοθεσία, κάνουμε διαβουλεύσεις πριν να κάνουμε οποιοδήποτε πρόταση, αυτό έγινε στα πλαίσια της Επιτροπής Γιούρκη και η διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να πω ότι τα τελευταία αυτά χρόνια έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και έχει αλλάξει κυρίως στους τομείς που ανέφερα και πρόκειται τώρα για συνήθι διαδικασία που ακολουθείτε στα πλαίσια της νομοθεσίας της εσείς είστε συνομοθέτε με το Συμβούλιο. Εσεί εγκρίνετε τις προτάσεις μας και τις κάνετε νομοθεσία και βεβαίω το Συμβούλιο χρειάζεται ενισχυμένη πλειοψηφία. Αντίθετα με το παρελθόν που χρειαζόταν η ομοφωνία αλλά δυσκόλευε τα πράγματα. Βεβαίω, υπάρχουν ακόμη κάποιοι τομείς στους οποίους αυτή η συνήθι διαδικασία δεν εφαρμόζεται. Και ξέρετε ότι υπάρχουν ακόμη ε, τομεί στου οποίου χρειάζεται ομοφωνία, επαναλαμβάνω. Για να μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση, πρότεινε η Επιτροπή η Πασχέλ, μια γέφυρα που ενώνει για να μπορέσουμε να μειώσουμε τα χάσματα που μας επιτρέπει να μπορούμε να, προχωρήσουμε, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ενισχυμένη πλειοψηφία. Και όλα αυτά υπάρχουν σε ένα έγγραφο και ελπίζω ότι θα ασχοληθείτε με τα θέματα αυτές. Τα τελευταία πέντε χρόνια και υπό την προεδρία του κυρίου Γιούνκερ και υπό την κυρία Τάισεν 27 νομοθετικές προτάσεις υποβάλαμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως για να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε τον πυλώνα και για να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα τριπλό α, όχι μόνο για τις τράπεζες αυτή τη φορά, αλλά και για την κοινωνική προστασία. Οι 24 από τις 27 αυτές προτάσεις έχουν ήδη εγκριθεί χάρη στη δική σας συμβολή πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές και εκκρεμούν ακόμα τρία νομοθετήματα, τα οποία βρίσκονται και στη μερίσια διαταξή σα. Ο νέο κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Το φθινόπωρο θα ξεκινήσουν τριμερεί διάλογοι για τα δύο αυτά νομοθετήματα και έχουμε και τον κανονισμό 883 για τον οποίο δυστυχώς δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε συμφωνία και για το οποίο θα σας μιλήσει η Επίτροπος Τάισεν λίγο αργότερα σήμερα όσον αφορά το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Τώρα, έχουμε καταφέρει να πετύχουμε νέους κανόνες όσον αφορά την ε, εξορρόπηση επαγγελματική και προσωπική ζωή. Νέοι κανόνε για την προστασία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια νέα πράξη προσβασιμότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου βασικά αγαθά και υπηρεσίε να είναι προσβάσιμα στα άτομα με ειδικέ ανάγκε, βελτιώντα κατά αυτόν τον τρόπο τη ζωή πάνω από 8 εκατομμύρια ανθρώπων. Έχουμε 26 χημικές ουσίες οι οποίες έχουν εντοπιστεί ως υπεύθυνε για την πρόκληση καρκίνου και για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έθεσε ανώτατα όρια έκθεσης. Αυτό το κάνανε οι συνάδελφοί μου που βρίσκονται στο Λουξεμβούργο. Αυτοί ασχολήθηκαν με το ζήτημα αυτό Συντοποιούμε ότι εδώ πέρα έγινε μια τεράστια νομοθετική εργασία και επιβάλλονται αυτή τη στιγμή πολύ σημαντικά πρόστιμα προκειμένου να προστατευτούν οι χιλιάδε αυτοί οι εργαζόμενοι οι οποίοι καθημερινά μέσω τη εργασία του εκτίθενται στι χημικέ αυτέ ουσίε. Επίση, μια σύσταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίθηκε όσον αφορά την κοινωνική προστασία και την προστασία στην εργασία. Έχουμε την εγγύηση για του νέου την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς επίσης και το νέο θεματολόγιο για τις δεξιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένες δεξιότητες και την επαγγελματική κατάρτιση, περιορισμένες εδώ είναι οι δυνατότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε ότι η εκπαίδευση παιδεία αποτελεί αντικείμενο εθνικής αρμοδιότητας. Όσον αφορά όμω την επαγγελματική κατάρτιση και τις σχετικές δεξιότητες, υπάρχουν αρμοδιότητες οι οποίες μπορούν να ληφθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αναλάβει και εμείς στην ουσιακό επίπεδο επίπεδο πολλέ δραστηριότητε για να βελτιώσουμε το υφιστάμενο σύστημα. Και αναφέρομαι σε αυτό που είπατε πριν από λίγο και εσεί, κυρία Πρόεδρε, πόσο σημαντικό να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργεια των νέων μέσω τη προώθηση των δεξιοτήτων. Το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει ασχοληθεί με αυτό και η επίτροπο Τάισεν, η οποία έχει επενδύσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού της κεφαλαίου προκειμένου να καταφέρει να προωθήσει περισσότερο την επαγγελματική κατάρτιση και προκειμένου να βελτιώσει αν θέλετε και την υπόλοιψη της κατάρτισης αυτής έτσι ώστε να μην επιθυμούν όλοι οι γονεί να στείλουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο προκειμένου να ακολουθήσουν μια θεωρητική κατάρτιση και εκπαίδευση, αλλά να μπορούν επίσης να επιλέγουν συνειδητά να στείλουν τα παιδιά του και σε προγράμματα επαγγελματική τεχνική κατάρτιση. Και επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι έχει εγκριθεί μια πολύ σημαντική νομοθεσία τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την προστασία των εργαζόμενων. Και θα ήθελα να μιλήσω τώρα στα γερμανικά. Η ελευθερία κίνησης ε, των εργαζομένων είναι μια θεμελιώδης ε, αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή τη στιγμή 17,5 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν καθημερινά αυτό το δικαίωμα και ζουν σε μία χώρα και δουλεύουν σε μία άλλη. Συνολικά, στην πατρίδα μου, ε, την Ολλανδία, έχουμε λίγο πολύ τον ίδιο πληθυσμό. Με την ε, επεξεργασία της οδηγίας για τους αποσπασμένους ε, εργαζόμενους ε, ε, θα εκπληρωθεί και η υπόσχεση του Προέδρου Γιούγκερ. Οι άνθρωποι που έχουν την ίδια εργασία να λαμβάνουν την ίδια αμοιβή. Για τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή ε, το 30 Ιουλίου του 2020 είναι η προθεσμία ε, βάσει αυτής ε, της οδηγίας και αυτή τη στιγμή έχουμε καλύτερη, καλύτερους κανονισμούς για την απάτη και για τους εργαζόμενους αλλά και για τους εργοδότες. Ξεκινά λοιπόν μια νέα φάση για την δίκαιη ρύθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Ε, επίσης έχουμε το έλεγχο στη Βρατισλάβα φέτος ε, ε, που θα πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το 2024 θα υποστηρίσει την ελευθερία κίνησης των εργαζομένων, την απόσπαση, θα υπάρχει ένα συντονισμός για την ασφάλεια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ε, για, κατά τις διαπραγματεύσεις για το ΕΛΑ, ε, το οποίο θα ψηφιστεί μέσα στο έτος. Θα συνεχίσω στα αγγλικά. Το δεύτερο μπλοκ, που είναι πιο σύντομο, το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Η δεύτερη βασική ε, ο δεύτερος βασικό τομέας εργασίας είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Είναι ο ετήσιος κύκλος οικονομικής και πολιτικής ε, μορφής συντονισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι νομοθεσία, είναι συντονισμός των εθνικών πολιτικών. Ο συντονισμός σε αυτό το εξάμεινο βοήθησε τα κράτη-μέλη να μεταρρυθμίσουν τα συστήματά τους και να επιστρέψουν στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και να μειώσουν τα επίπεδα ανεργίας στις ε, επικράτειές τους. Έχουμε κυκλοφορήσει ένα φύση, ένα δελτίο, ε, το, το Σεπτέμβριο του 2019 θα δείτε από τις διαφάνειες που περιλαμβάνει πόσο έχουν πέσει τα ποσοστά ανεργίας και ότι συνεχίζουν να πέφτουν. Φυσικά όλα αυτά ε, συγκρίνονται και με το βάθος της κρίσης. Πρέπει δηλαδή να μην ε, υπάρχει εντύπωση ότι αυτές τις δουλειές τις έφτιαξε η Κομισιόν. Ήταν οι επιχειρήσεις, τα κράτη-μέλη ε, που έφτιαξαν αυτές τις θέσεις Επίσης ε, έχουμε και τον ε, μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάντοτε ως γραμμή βάσης είναι η κρίση. Τα πάντα λοιπόν συγκρίνονται με αυτή τη λυπηρή κατάσταση και είναι μέση όρη. Και αν δείτε το μέσο όρο κράτος μέλος, θα έχετε μεν μία εικόνα, αλλά αν πάτε με λεπτομέρεια στην κάθε περιφέρεια μπορείτε να δείτε ε, μια πολύ διαφορετική εικόνα, περιοχές με πολύ υψηλή ανεργία που είναι απομονωμένες κτλ. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι από τότε που ξεκίνησαν αυτές οι στατιστικές ποτέ δεν είχαμε τόσους πολλούς εργαζόμενους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται επίσης ότι η εργασία των γυναικών αυξάνεται κάθε χρόνο και αυτή είναι η στόχη που εμείς οι ίδιοι θέσαμε. Βέβαια όχι όλοι οι πολίτες και όχι όλες οι χώρες ε, με τον ίδιο τρόπο. υπάρχουν κάποιες ε, κατηγορίες ε, ε, τα παιδιά, οι νέοι, τα άτομα με αναπηρία, οι εθνικές μειονότητες, όπως η Ρώμα, χρειάζονται συνεχώς προστασία. Και βέβαια πρέπει να κάνουμε κάτι για τους αστέγους και να δώσουμε και πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες. Ένα σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξή μας. Το ευρωπαϊκό εξάμεινο γίνεται όλο και πιο κοινωνικό θα έλεγα. Ε, πάει σε τομείς ε, που είναι πέραν των κλασικών τομέων όπως είναι αυτοί με τους οποίους ασχολείται το Υπουργείο Οικονομικών. Το βασικό μήνυμα που θέλω να σας δώσω σήμερα είναι ότι πρέπει να το λάβετε στα σοβαρά υπόψη. Δεν είναι ε, κάτι, ένα εργαλείο το οποίο αφορά μόνο τους υπουργούς οικονομικών. Έχει ένα πολύ ισχυρό κοινωνικό κομμάτι. Ο Γιούγκερ και η Τάισεν έχουν πολύ εργαστεί ε, ε αυτού του θέματος. Έχουμε το κοινωνικό scoreboard που συγκρίνονται τα κράτη-μέλη βάσει συγκεκριμένων συγκρίσιμων κριτηρίων. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, ε, γιατί με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να πάρουν μέτρα για να μην βρίσκονται ουραγοί και υπάρχουν και τα CSRs, ε, οι συστάσεις αναχώρα και οι αποφάσεις που παίρνει το Συμβούλιο και όχι η Κομισιόν ε, που συστήνουν στα κράτη-μέλη να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Θα δείτε και εκεί την κοινωνική διάσταση. 45% όλων των συστάσεων, αν δείτε στο παρελθόν, ήταν για κοινωνικά θέματα και για τις δεξιότητες. Άλλη μια φορά οι δεξιότητες. Επίσης, η νέα πρόεδρος της Κομισιόν έχει αποφανθεί υπέρ αυτής της διαδικασίας και ήταν πολύ πιο ξεκάθαρη. Δηλαδή, μας ζήτησε να ερχόμαστε και να συζητάμε με το Κοινοβούλιο πριν από κάθε νέο βήμα στη διαδικασία του εξαμήνου. Το τρίτο μπλοκ είναι τα κονδύλια, όπως είπα. Το πιο σημαντικό είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που είναι και στη συνθήκη. Πάνω από 16 χρόνια, 60 χρόνια ήταν το βασικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, για την επόμενη περίοδο 21-27 η Κομισιόν προτείνει να γίνει ακόμα πιο ισχυρό και θα ονομάζεται Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ, ESF+. Η ε, ε, Κομισιόν έχει προτείνει προτείνει ένα ταμείο με 101,2 δις ευρώ για 7 έτη, που είναι λίγο πολύ το ίδιο ποσό με αυτό που διαθέτουμε σήμερα, αν το μετρήσετε σε πραγματικά χρήματα. Είναι μια πολύ σοβαρή δέσμευση, αν δείτε γενικά πόσο υποπίεση βρίσκεται ο προϋπολογισμός και δεν θέλω να αναφέρω και τις επιπτώσεις του Brexit. Άρα αυτό μεταφράζει ακριβώς ε, την αξία που δίνει η Κομισιόν στην κοινωνική Ευρώπη και είναι και το 1 δέκατο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Γιατί ονομάζεται ESF+. Γιατί σε ένα νομικό κείμενο συνδυάζουμε τέσσερα διαφορετικά ταμεία. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά και τέσσερα άλλα που σήμερα έχουν δικό τους ε, κανονισμό. Έτσι λοιπόν δημιουργούμε καλύτερες συνέργειες ε, και ευθυγραμμίζουμε τις διαδικασίες. Ε, υπάρχει ε, για το ΓΕΙ, για το ε, ΦΕΑΝΤ και για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κοινωνικής Καινοτομίας, το EASY όπως το λέμε εμείς, και υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Υγείας που δεν νομίζω ότι είναι στη δική σας επιτροπή, στη δική σας αρμοδιότητα, όμως θα εντάσσεται στο ESF Plus στο μέλλον με μια πιο αξορθολογισμένη διαδικασία διαχείρισης. Επίσης υπάρχει το EGF που επεμβαίνει μετά από ε, ένα συμβάν. Το ESF είναι το εργαλείο που βοηθά τα κράτη-μέλη να προβλέπουν, να εξυγχρονίζουν τις αγορές εργασίας, να κάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την παγκοσμιοποίηση έρχεται μετά, εκ των υστέρων, για τους ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά τους λόγω της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Εμείς λοιπόν ε, ζητάμε τη δική σας βοήθεια και συνδρομή και ε, στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Σήμερα έχουμε και το ε, Juncker Fund, το οποίο στο μέλλον θα ονομάζεται Investing EU, που είναι δάνεια. Στην προηγούμενη περίπτωση είχαμε χορηγήσεις, ενώ στο Investing You έχουμε δάνεια, τα οποία δίνονται από τις τράπεζες με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε και ένα κοινωνικό παράθυρο 4 δις ευρώ που θα κινητοποιήσει περίπου 50 δις μέσα από την μόχλευση επενδύσεων. Είναι μια πολύ σημαντική νέα πρόταση λοιπόν και τέλος ο κοινωνικός διάλογος. Να αναφέρω βέβαια ότι είναι κέρια σημασίας. Η Κομισιόν αυτή θα δώσει νέα πνοή στον κοινωνικό διάλογο. Θέλει να ενισχύσει το ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και σε εθνικό επίπεδο. Η Γενική Διεύθυνση επίσης είναι υπεύθυνη για τον διάλογο ε, μεταξύ των διαφορών κλάδων, ε, σε κλαδικό δηλαδή επίπεδο και σε τομεακό επίπεδο. Και επίσης ε, είμαστε, έχουμε αφοσιωθεί και στην σωστή λειτουργία του κοινωνικού διαλόγου. Υπάρχει η τριμερής ε, κοινωνική σύνοδος κορυφής που θα δώσει επίσης μια νέα διάσταση στο θέμα. Τέλος, να πω δεν θέλω να πω ότι η κοινωνική εταίρεια είναι το ίδιο με την κοινωνία των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει είναι σημαντική για μεγάλο κομμάτι των πολιτικών μας. Ε, αυτά είχα να πω για τα βασικά στοιχεία της δράσης της Γενικής Διεύθυνσής μας. Ίσως να μακρηγόρησα, όμως ήθελα να πω και κάποια πράγματα για το μέλλον. Τι θα γίνει στο μέλλον. Βέβαια, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή να επισκιάσω τι κατευθύντηρε γραμμέ τη νεοκλεγή σα Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στι οποίε είδατε κάποιε πολύ σημαντικέ πρωτοβουλίε. Περισσότερε πρωτοβουλίε θα δούμε και τι υπόλοιπε 100 μέρε. Βέβαια, Εμεί, από τη δικιά μου τη Γενική Διεύθυνση, καθώ επίση και οι συναδελφοί μου από τις υπόλοιπε Γενικές διευθύνσει ακολουθούμε συγκεκριμένου πολιτικούς κανόνες και πολιτικούς προσανατολισμού, Πρέπει να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα. Αυτή τη στιγμή αρχή συνεργάζεται η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει αυτή τη στιγμή βέβαια να είμαι πάρα πολύ προσεκτικό επισερχόμενο σε περισσότερες λεπτομέρειες και σε κάθε περίπτωση εκφράζουμε υπό την επίβλεψη της κυρίας Τάισεν. Και σαφώς δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας δώσω απόλυτες εγγύσεις για το τι μελιγενέστε με την Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την 1η Νοεμβρίου και μετά. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα ήθελα να κάνω τις εξή παρατηρήσεις. Σε σχέση με το που βρισκόμασταν το 2014-2015 η κατάσταση έχει σαφώς βελτιωθεί. Το κοινωνικό καθεστώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εν γέννη βελτιωθεί. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εφησυχάσουμε. Έχετε δει τα αριθμητικά δεδομένα, κινούνται σε σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να επαναπαυτούμε σε καμία περίπτωση, το αντίθετο μάλιστα. Ήδη σα είπα ότι υπάρχουν ακόμα πολύ μεγάλε αποκλήσει και ανισότητε μεταξύ των κρατών μελών, πολύ σημαντικοί θύλακες ένδια και φτώχεια σε ορισμένα κράτη-μέλη και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με εσά, με τα κράτη-μέλη, με του κοινωνικού εταίρου. Έχουμε μειονεκτούσε ομάδε στις οποίε αναφέρθηκα, τι οποίε θα πρέπει να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ και στο μέλλον και έπειτα έχουμε και τι γενικότερε αναδυόμενε τάσει, εμφανίσει σε όλου, και οι οποίες θα απαιτήσουν σε ορισμένες περιπτώσεις να αναθεωρήσουμε κάπως ε, τα μοντέλα τα οποία ακολουθούμε το μέλλον της εργασίας, το μέλλον της απασχόλησης για παράδειγμα. Αυτό θα πρέπει να σε απασχολήσει. Νέες μορφές συμβάσεων, λιγότερες συμβάσεις ενδεχομένω, πιο επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. Πώς μπορούμε λοιπόν να προσαρμόσουμε το σύστημά μας, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν το σύστημα απασχόληση, πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τι δημογραφικέ τάσει οι οποίε συναντίονται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όλα αυτά απαιτείται περαιτέρω πολιτική δράση τα επόμενα χρόνια. Και έπειτα έχουμε και το ζήτημα του μετασχηματισμού, της μετάβασης. Μετάβαση και μετασχηματισμός εξαιτία της κλιματικής αλλαγής. Το 2050 θα πρέπει να έχουμε φτάσει σε μια οικονομία οποία θα είναι ουδέτερη ως προς την κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε όμως και στην τεχνητή νοημοσύνη. Πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε εν γέννη τις κοινωνίες μας χωρίς να χάσουμε το πολύτιμο μοντέλο απασχόλησης το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα αυτό και αν διαβάσετε εκ νέου το λόγο της νεοκλεγής Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δείτε ότι επικεντρώνεται πάρα πολύ στο ζήτημα αυτό. Εγώ θα ήθελα πολύ να εστιαστώ σε αυτό το ζήτημα και θα το καταφέρω βέβαια μόνο αν έχω τη δική σας την υποστήριξη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εμεί σας ευχαριστούμε κύριε Κόρτε για την παρουσία σας αυτή. Θα δώσω το λόγο καταρχάς στους συντονιστές μας. Πιέζει όμως πολύ ο χρόνος. Θα σας ζητήσω λοιπόν να τηρήσετε το χρόνο αγόρευσης δύο λεπτά ο καθένας προκειμένου να κάνετε παρατηρήσεις, να θέσετε ερωτήσεις. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο κύριος Ράτικ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Κόρτε. είδαμε στην ουσία τις επιτυχίες της τελευταίας νομοθετικής περίοδου. Είδαμε όμως δυστυχώς και στην εκλογική αναμέτρηση πόσο σημαντικό ε, είναι ο ρόλος που παίζει στο μυαλό των ανθρώπων το κοινωνικό κομμάτι. Κανένας. Ε, θα πρέπει λοιπόν μάλλον να προχωρήσουμε με πιο θετικό τρόπο έτσι ώστε οι άνθρωποι να αρχίσουν να εποφελούνται από αυτές ε, τις επιτυχίες που αναφέρατε και να μην παραμένουν τα όσα είπατε μεταξύ μας. Έχουμε ήδη μιλήσει για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Είπατε ότι είναι κοινωνικό εξάμεινο, κάτι που μου λείπει πολύ επίσης κοιτώντα ε, το social scoreboard, ε, το θέμα των διαπραγματεύσεων για τους μισθούς. Μιλήσαμε για το ευρωπαϊκό ελάχιστο μισθό. Ε, υπάρχουν τέτοιες αναφορές όμως τελικά στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμείς έχουμε την κοινωνική αγορά εργασίας και ε, ο ελάχιστος μισθός είναι απλώς ε, μία ε, πατερίτσα. Εμείς θέλουμε κοινωνικό διάλογο, συλλογικές διαπραγματεύσεις, ώστε να μην υπάρχει πολιτική ασυδοσία. Θέλουμε ε, να δούμε πώς ακριβώς διαμορφώνεται το σύστημα με τους μισθούς στα κράτη-μέλη και να επικεντρωνόμαστε στην την Ευρωπαϊκή Αρχή της Κοινωνικής Οικονομίας που είναι πολύ σημαντική για εμάς. Ευχαριστώ κυρία Γιουγκέριος για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κόρτε για την παρουσίαση της Γενικής Διεύθυνσης ΕΜΠΛ και της δουλειάς που έχει γίνει. Νομίζω ότι ότι σωστά ξεκινήσατε με τον Ευρωπαϊκό Πυλόν των Κοινωνικών Δικαιωμάτων ως βάση αρχών και μιλήσατε και για πολιτική δέσμευση. Αυτή η κοινή πολιτική δέσμευση είναι που με απασχολεί. Γιατί ακούμε που και που τις ομιλίες ε, της νέας Προέδρου της Επιτροπής αλλά με, ακούγοντας τις υποσχέσεις της, πραγματικά αναρωτιόμαστε πώς θα εφαρμοστούν αυτές οι υποσχέσεις. Μιλήσατε για το ε, ένα δίκαιο ενίκιο που μπορεί κανείς να πληρώσει, αυτό είναι ένας ε, από τους στόχους. Θα αυξηθούν ενδεχομένως τα σπίτια που θα μπορεί κανείς να νοικιάσει με ένα ε, χαμηλό ποσό. Όμως δεν είναι μεγάλος και ο κίνδυνος λόγω της επικουρικότητας να ρίξουμε την ευθύνη στα κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν τις υποσχέσεις του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Άρα, συγκεκριμένη ερώτηση. Πότε θα καταθέσει η Κομισιόν μια συγκεκριμένη πρόταση, γιατί μιλήσατε για την επισφαλή εργασία και το μέλλον της εργασίας και οι άνθρωποι στην... Οι άνθρωποι που δουλεύουν σε πλατφόρμες ε, που έχουν προβλήματα γιατί οι πλατφόρμες θεωρούν ότι δεν είναι υπεύθυνοι για τις ε, εργασιακές σχέσεις είναι σε δύσκολη θέση. Φαίνεται λοιπόν ότι χρειάζεται μια τέτοια πρόταση για δίκαιες συνθήκες εργασίας, ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους. Ο κύριος Μησινάρου Θα ζητήσω από την συνσυντονιστριά μου στην ομάδα Renew να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Συντονιστά, κυρία Πρόεδρε και Γενική Διευθυντή για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη. Στην ομάδα μας επιμένουμε στην εφαρμογή ε, του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Υπάρχει ε, ανάγκη να βασιστούμε σε αυτό, ειδικά όσον αφορά ε, στα τρία τελευταία στοιχεία που αναφέρεται, το ESF+, το EGF, ε, θα χρειαστούμε σίγουρα ε, αυτά τα ε, ταμεία τους επόμενους μήνες και επίσης συντονισμός για τον κανονισμό 883. Τα άλλα σημαντικά θέματα στη δική μας ομάδα είναι να συνεχίσουμε ε, στον δρόμο της μείωσης της ανεργίας των νέων, ειδικά των νέων που είναι η λεγόμενοι νέτ, δεν είναι ούτε σε εργασία, ούτε σε εκπαίδευση. Θέλουμε να ενισχύσουμε την ε, νεολαία μας και τέλος όσον αφορά την ε, προετοιμασία για τη μετάβαση, όσον αφορά τις δεξιότητες, την εκπαίδευση, ε, την οικονομική μεταμόρφωση και μεταρρύθμιση, είπατε ότι συνεχώς οι εξελίξεις επιταχύνονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ε, η οικονομία αλλάζει, οι δεξιότητες που απαιτούνται αλλάζουν, αλλά υπάρχει και το οικολογικό κομμάτι, η οικολογική διάσταση. Μιλάμε για, τις, ε, ε, τα, για αυτά που χρειάζονται σε περιβαλλοντικό επίπεδο να δω, μπουν ανώτατα όρια έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις τάσεις που τόσο πολύ ε, φοβούνται οι άνθρωποι. Χρειάζεται το μίνιμουμ λοιπόν για να εφαρμόσουμε αυτά που θέλουμε. Τώρα εκ μέρους των Πρασίνων η κυρία Λάγκεν Ζίμπεν. Ευχαριστώ κύριε Κόρτε. Θα αναφέρω κι εγώ κάποια στοιχεία ε, σχετικά με τη, όσα θέλει η δική μας ομάδα. Ευχαριστώ πολύ για τα όσα αναφέρετε. Όμως νερώνουμε το κρασί μας, ε, γιατί στο μεταξύ υπάρχουν ε, πάρα πολύ σημαντικοί ε, νόμοι οι οποίοι αναβάλλονται και δεν έρχονται τη στιγμή που θα τις θέλαμε. Ας πούμε, η οδηγία για το χρόνο εργασίας. Μιλήσατε για την υγεία να σας αναφέρω την οδηγία για τα μειοσκελετικά νοσήματα. Πριν από μερικές εβδομάδες στη Γερμανία είχαμε μια πολύ έτσι, ε, ζωηρή συζήτηση για προβλήματα ε, αναπνευστικά, όχι μόνο μειοσκελετικά. Μιλήσαμε λοιπόν για τα νοσηλευτικά ιδρύματα, πώς πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να αντιμετωπίζονται Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, έγινε λοιπόν μια συζήτηση και με τον Υπουργό ε, Υγείας. Αυτά είναι θέματα που καίνε. Ε, θέλουμε λοιπόν μια συγκεκριμένη οδηγία γιατί μας την έχουν υποσχεθεί και θα θέλαμε να συνεχιστεί η προσπάθεια και τα επόμενα χρόνια. Ε, ο ελάχιστος μισθός, πολύ σημαντικό θέμα, το χαιρετίζουμε χαιρόμαστε που θα υπάρχει μελλοντικά συνεργασία. Χρειαζόμαστε νόμους. Δεν χρειαζόμαστε συστάσεις από το Συμβούλιο. Θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα, να δούμε πού ακριβώς ε, χρειάζεται να δράσουμε για να γίνει ορατή η κοινωνική πολιτική για να μπορέσουμε να φέρουμε στους ανθρώπους στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Για την ταυτότητα και τη δημοκρατία η κυρία Ζόμε. Σας ευχαριστώ. Με μεγάλη προσοχή άκουσα τι είπατε, αλλά πρέπει να πω ότι κάποια θέματα με απασχολούν. Θα μιλήσω για αυτό το νέο ίδρυμα για την εργασία που θα γεννηθεί τον Οκτώβριο. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνει, τι, με ποια θέματα θα ασχοληθεί όσον αφορά το κοινωνικό dumping τι γίνεται. Πρέπει να πω ότι εμείς έχουμε στις ε, διάφορες περιοχές της ε, χώρας μου διάφορα γραφεία τα οποία προμηθεύουν εργαζόμενους οι οποίοι έχουν αποσπαστεί από κάπου και πολλού να εργαστούν σε εμά. Τι γίνεται λοιπόν. Πρέπει να πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει, ε, είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά τα κυρίαρχα δικαιώματα των εργαζομένων. Τι θα κάνει αυτός ο οργανισμός. Επίσης, θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον δεν θα έχει τέτοιου είδους προνόμια που να μπορεί κατά κάποιο τρόπο να υπερέχει των εθνικών ρυθμιστικών οργάνων και να επιδεινώσει τα κοινωνική προστασία των εργαζομένων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόκκινγκ για το ECR. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή και αυτή την ε, ανάλυση που ήταν ιδιαίτερα μακροσκελής. Ε, κατανοήσαμε ότι μελλοντικά στην Ευρώπη θα έχουμε ζητήματα για, με, λόγω της κλιματικής αλλαγής, ε, λόγω της ανέχειας, της ανεργίας των νέων. Αυτές είναι οι λέξεις κλειδιά. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρόνια που έχουμε μπροστά μας για να μπορέσει να προσαρμοστεί η οικονομία της Ευρώπης και να διαμορφωθεί κοινωνικά η Ευρώπη, να νιώσουν οι άνθρωποι την Ευρώπη, ε, να, να δείξουμε ακριβώς ε, ότι πάμε στη ρίζα του ευρωπαϊκού πολιτισμού που είναι η οικογένεια και νομίζω ότι έχουν, ε, έχει έρθει η στιγμή για μια μεγάλη συζήτηση για να μπορέσουμε να ενεργοποιηθούμε ώστε να νιώσει ο κόσμος στην Ευρώπη έτσι ώστε συγκεκριμένες, ε, συγκεκριμένα μορφώματα να μην βρίσκουν ε, πρόσφορα έδαφος. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας. Είναι 4-5 χρόνια που χρειαζόμαστε γι' αυτό. Αν δεν γίνει θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Έχουμε πολλά ε, πράγματα αποφασίσει. Έχουμε επίσης διαγράψει κάποιες δράσεις για να γίνουν εξοικονομήσεις χρημάτων. Όμως ε, ε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα κοινωνικά project για να έχουμε ένα ε, καλύτερο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την ανάλυση σας και για τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ. Now, give the floor to τώρα θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις. Συγγνώμη, συγγνώμη, ξέχασα την ΚΟΕ, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Κύριος Βίλιονσεν. Ευχαριστώ. Δεν καλό να μας ξεχνάτε, διότι είμαστε μια σημαντική πολιτική ομάδα. Και αν μας ξεχνάτε θα είμαστε εδώ να σας το υπονθυμίζουμε. Σας ευχαριστώ που δώσετε το λόγο, σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ κύριε Γενική Διευθυντά. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο διάλογος. Θα ήθελα να ερωτήσω το εξής. Σε σχέση με την επιδημία της κυρίας Φαντελάιν, να εισαγάγει την έννοια αυτού του σε κατώτατης ευρωπαϊκής αμοιβή. Νομίζω ότι θα πρέπει πρόταση αυτή να γίνει τις πρώτες 100 ημέρες. Θα ήθελα να σας ερωτήσω, ποια είναι η γνώμη σας, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το μέσο ευρωπαϊκό όρο, το ποσό θα είναι το ίδιο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει σεβαστό αυτό. Κυρίως αριστερά από τις ε, σκανδιναβικές ε, χώρες, όπου όλα αυτά τα θέματα δεν αποφασίζονται από την νομοθεσία, αλλά είναι αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμφωνίες μεταξύ όλων των κοινωνικών εταίρων. κύριος Χόσκιν. Βλέπω ότι ο κύριος ε, Χόσκιν μιλά πολύ καλά πολλές γλώσσες. Θα μιλήσω τσέχικα. Ίσως αργότερα. Να δω αν γνωρίζει επίσης και τσέχικα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κόρτε. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ πρέπει να πω ότι επισκέφθηκα τον οργανισμό που είναι υπεύθυνο με θέματα διαχείρισης απασχόλησης ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Είπαν ότι έχουν καλά αποτελέσματα μέχρι τώρα, αλλά κατά πόσον έχει μέλλον. Λαμβάνεται υπόψη τα αποτελέσματα ε, των μελετών που κάνει. Θα πρέπει να σκεφτούμε αν αυτός ο οργανισμός δεν θα έπρεπε λίγο να αλλάξει, να μεταρρυθμιστεί. Όσον αφορά τις κοινωνικές ανισότητες σε κάποιες χώρες, η Αυστρία για τους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει μείωση των επιδομάτων και βοήθειας που δίδεται για τα ανήλικα άτομα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο κριτικής. Μας απασχολεί όμως εμάς τι θα κάνει στα πλαίσια αυτού του θέματος Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τον προπολογισμό, πιστεύετε ότι έχουμε αρκετά θετικά project και σχέδια. Εδώ αποδεικνύεται ότι τα τελευταία χρόνια οι πολιτικές και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πολύ θετικά, αλλά θα πρέπει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να αλλάξουμε, να βελτιώσουμε τα πράγματα και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα διαθέσιμα κονδύλια με τρόπο πιο αποδοτικό. Ευχαριστώ. Κύριος Ντάνιελσον, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω σου ειδικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το Γενικό Διευθυντή για την παρουσίαση που έκανε. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι ε, ακούσαμε ότι μέσα σε επόμενες 100 μέρες θα έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις ελάχιστες αποδοχές, τον λεγόμενο ελάχιστο μισθό. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, ιδίω για τους κοινωνικούς εταίρους. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα πολλά διαφορετικά πρότυπα και μοντέλα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαμόρφωση του λεγόμενου ελάχιστου κατώτατου μισθού. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν 4.000 άνθρωποι οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της εργασίας. 80.000 χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας της έκθεσης σε επικίνδυνη ακτινοβολία. Και υπάρχουν βέβαια και πολλά κοινωνικά, ψυχολογικά προβλήματα τα οποία προκύπτουν στο χώρο εργασίας και τα οποία έχουν δυσμενέστατες καταστροφικές συνέπειες για τις ζωές των Ευρωπαίων πολιτών. Νομίζω λοιπόν ότι στα πλαίσια της στρατηγικής για την απασχόληση που θα καταρτήσετε θα πρέπει να έχετε και μια τέτοια φιλοδοξία ουσία. Μηδενικά εργατικά ατυχήματα. Μηδενική εργατική θάνατη για του εργαζομένου. Όσοι σηκώνται το πρωί για να πάνε στη δουλειά θα πρέπει να μπορούν να επιστρέφουν το βράδυ στο σπίτι του. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει εδώ πέρα να κάνετε μια συγκεκριμένη πρόταση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρησιμοποιώντα όμω και συγκεκριμένου δείκτε και αριθμητικά δεδομένα τα οποία μπορεί να συλλέξετε από τι αρμόδιε αρχέ των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε ειλικρινά να έχουμε ένα πιο φιλόδοξο πρόγραμμα για τη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να έχουμε πραγματικά ένα στόχο μηδενικό όσον αφορά τους θανάτου και τα ατυχήματα. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μάντερς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκπροσωπώ τους εργαζομένους άνω των 50 από τις κάτω χώρες Αναφερθήκαμε πριν από λίγο στην ε, προεκλογική εκστρατεία, στις υποσχέσεις που δόθηκαν. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σαφώς προωθεί την ευημερία, την οικονομική, αλλά Πολύ συχνά στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλούσε μόνο για τι μεγάλε πολυεθνικές επιχειρήσει. Α καλύψουμε πλέον και του ανθρώπου αυτού που βρίσκονται στη δυσχερή εκείνη κατάσταση να μην μπορούν να έχουν ένα ασφαλέ επαγγελματικό μέλλον. Και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα καταφέρουν να καταλήξουν σε μια λύση. πώ μπορούν να ενσωματώσουν τους αποκλεισμένους αυτούς ανθρώπου. Δεν μιλάμε μόνο για εισοδήματα και για μισθό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτό το κοινωνικό χάσμα όπως αποκαλείται να επανανταχθούν στην κοινωνία όχι μόνο μέσω αποδοχών και χρημάτων αλλά να μπορούν να προστατεύονται από κοινωνικής πλευράς σε καθημερινό επίπεδο, να ενταχθούν σε ένα νέο κοινωνικό πλαίσιο. Σας Προκαλώ λοιπόν να βρείτε μαζί με εμά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάποιες λύσεις... και για του ανθρώπους εκείνους, τους πιο ηλικιωμένου οι οποίοι αποκλείονται από την ε, κοινωνία τους όχι μόνο σε ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά γενικά αποκλείονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα. Ελπίζω ότι θα αποδεχθείτε την πρόκλησή μου αυτή και ότι θα καταφέρουμε τα επόμενα χρόνια να καταλήξουμε από κοινού σε μία λύση προκειμένου να επανεντάξουμε τους ανθρώπους αυτούς στην κοινωνία, όχι μόνο από οικονομικής αλλά και από κοινωνικής κυρίως πλευρά. Σας ευχαριστώ. ο κύριος Σαλίμπα και ο κύριος, και ο στη συνέχεια. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Κόρτε, για τη λεπτομερέστατη παρουσίαση που μας έκανε. Δύο ερωτήσει θα ήθελα να θέσω. Πρώτον, όσον αφορά τα επικείμενα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πολύ συχνά στο παρελθόν ακούσαμε να γίνεται λόγος για την ψηφιοποίηση. Ψηφιοποίηση Τη απασχόληση του χώρου εργασία και ποιε είναι οι επιπτώσεις που μια τέτοια ψηφιοποίηση μπορεί να έχει ή ήδη έχει για τους Ευρωπαίους εργαζομένους. Νομίζω ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αρχίσει να επεξεργάζεται νομοθετικές προτάσεις για να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις που η ψηφιοποίηση μπορεί να έχει στο χώρο εργασίας. Το δικαίωμα της ηλεκτρονικής ψηφιακής αποσύνδεσης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έχει ήδη απασχολήσει κράτη-μέλη η Γαλλία όπου βλέπουμε ότι εκεί έχουμε θετικές επιπτώσεις από τον νόμο που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται στη χώρα αυτή. Διερωτάμε λοιπόν στο νέο πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν κάποια σχετικά δικά σας σχέδια προκειμένου να καλύπτεται και το δικαίωμα αυτό της ψηφιακής αποσύνδεσης και προκειμένου να ισχύει παντού σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή. Όσον αφορά τώρα την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, εγώ θεωρώ ότι το Ταμείο αυτό θα πρέπει να καλύπτει όλες τι πραγματικότητε, ακόμα και εκείνες που αντιμετωπίζουν τα μικρότερα κράτη-μέλη, όπως η Μάλτα. Στη Μάλτα, τη δική μου τη χώρα, δεν έχουμε πολλές επιχειρήσεις που να απασχολούν πάνω από 500 εργαζόμενους. Προκειμένου λοιπόν να καταφέρουμε να μπορούμε να αποφεληθούμε και εμείς κατά τρόπο αποτελεσματικό από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει απαραίτητη μεταρρύθμιση του ταμείου αυτού προκειμένου να μπορεί να καλύπτει και την κατάσταση εκείνη στην οποία βρίσκονται κρατημέλη όπως όπω η Μάλτα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε έχουν και μικρότερες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερου εργαζόμενους. Και νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να μειωθεί εν γέννη ο αριθμός των ανέργων. Ας ακούσουμε την επόμενη ομιλητή και στη συνέχεια την κυρία Μπλικενβιτσούτε. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ ότι ε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση που μας έκανε ο Γενικό Διευθυντή. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να πούμε κάτι πάρα πολύ απλό και σαφές αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο του κοινωνικού πυλώνα διακυβεύεται το μέλλον της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο το μέλλον των κοινωνικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διακυβεύεται το ίδιο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούμε όντω την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, τα θετικά αποτελέσματα που έχουμε εδώ και εκεί. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει ξεκάθαρα να πούμε ότι ως προς το κοινωνικό χάσμα, ως προς την κοινωνική ανισότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα και θεωρώ ότι αυτό είναι ο αδύνατος κρίκος αυτή τη στιγμή της πρόκλησης του στοιχήματος που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά δηλαδή την οικονομική και κοινωνική ευημερία θα ήθελα να αφαιρθώ σε τέσσερα σημεία. Ελάχιστε αποδοχέ, κατώτατο μισθό. Το ζήτημα αυτό προφανώ θα πρέπει να το συζητήσουμε με του κοινωνικού εταίρου και να δούμε πώ στην πράξη μπορεί να εφαρμοστεί μια τέτοια πρόταση. Και συμφωνώ εδώ πέρα με όλου του συναδέλφου οι οποίοι αναφέρθηκαν στο ζήτημα αυτό, που είπαν ότι θα πρέπει όντω επιγόντω το ζήτημα αυτό να αντιμετωπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ζήτημα τη στέγαση, κατά δεύτερο λόγο. Ποιε πολιτικέ για τη στέγαση θα έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτικέ οι οποίε να ισχύουν για όλου όμω του πολίτε. Νομίζω ότι και εδώ χρειαζόμαστε συγκεκριμένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να εμβαθύνετε λίγο περισσότερο, κύριε Γενική Διευθυντή. Τρίτον, το ζήτημα της περιθεωριοποίησης, τι, τι γίνεται με τους απόρους, με τους αστέγους. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δούμε ότι το ζήτημα των ανθρώπων αυτών συνδέεται με την αποτυχημένη απόπειρα ένταξης των μεταναστών. Και τέλος, τι πρόκειται να γίνει με τις πολιτικές που έχουν ως στόχο την τρίτη ηλικία, τους πιο ηλικιωμένους. Ξέρετε, εδώ πέρα πρέπει να δούμε δύο ξεχωριστές πτυχές του ζητήματος. Την ενεργή γύρανση του πληθυσμού δηλαδή πώς μπορούμε να στηρίξουμε τους εργαζόμενους ηλικιωμένου και έπειτα τι μπορούμε να κάνουμε με τους ανθρώπους εκείνους ηλικιωμένου οι οποίοι δεν μπορούν πλέον οι ίδιοι να φροντίσουν τον εαυτό τους, οι οποίοι δεν είναι αυτάρκες και αυτόνομοι. Νομίζω ότι και από αυτού του ζητήματος θα πρέπει να αναλυφθούν πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Μπλικεντζιτσούτ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γενική Διευθυντά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση που κάνετε, για τη συνεργασία που έχουμε και η γενική σας διεύθυνση πρέπει να πω ότι επιτέλεσε πολύ παραγωγικό έργο. 25 ε, νομοθετήματα από τα οποία 24 εγκρίθηκαν. Εγώ είμαι επί του στα θέματα της παγκοσμιοποίησης και πρέπει να πω ότι με πολύ ενεργό τρόπο θα συνεργαστούμε για να εγκριθεί το συντομότερο δυνατό το, η έκθεση αυτή, διότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό για τους πολίτες μας. Θα σας θέσω την εξής ερώτηση. Ο κοινωνικός πυλώνας είναι πολύ σημαντικός. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν αυτό το κοινωνικό πυλώνα. Εγκρίναμε τις 20 Γενικές Αρχές το 2017 και η ερώτησή μου είναι η εξή. Η Γενική σα Διεύθυνση θα αποτιμήσει τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ετών. Τι δεν έχει γίνει ακόμη, ποιες είναι οι προτεραιότητες, πώς θα τις ιεραρχήσουμε. Δεύτερη ερώτηση, ποια είναι η άποψή σας για τις ευρωπαϊκές εγγύησεις για τα παιδιά, κυρίως όσον αφορά την φτώχεια των παιδιών. Η σοσιαλιστική ομάδα έθεσε πολλές φορές το θέμα αυτό. Ποια είναι τα μέσα που διατίθενται για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια των παιδιών. Μέχρι τώρα τα μέσα είναι ανεπαρκή. Θα πρέπει λοιπόν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να συντονιστούμε για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το τρομερό πρόβλημα. Οι προτάσεις είναι καλές, οι συστάσεις επίσης καλές, αλλά για ποιο λόγο τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να θέσουν σε εφαρμογή αυτές τις συστάσεις. Πού είναι το πρόβλημα. Πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε τους στόχες μας. Ευχαριστώ. Ε, συνεχίζουμε με την κυρία Στάνοκα και η κυρία Χόμσκα παρακαλώ προετοιμαστείτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Κότς, θα ήθελα να αναφέρω τρεις προτάσεις που αναμένουμε ενδεχομένω. Πολλοί συνάδελφοι μέχρι τώρα ανέφεραν τον, την κατώτατη αμοιβή. Ένα άλλος ε, δείκτης που υπάρχει στις συστάσεις είναι το κατώτατο εισόδημα. Τι γίνεται με το θέμα αυτό. Δεύτερον, υπάρχει το θέμα της ε, προστασίας των εργαζομένων ε, στο χώρο εργασίας από διάφορες ασθένειες ενδεχομένως που μπορούν να προκαλούνται. Επίσης, αναμένουμε από την Επιτροπή την ε, οδηγία πλαίσιο για την συμμετοχή των εργαζομένων ε, σε θέματα κοινωνικά που τους ενδιαφέρουν. κυρία Χόμς και να προετοιμαστεί η κυρία Φράνσεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κόρτε που είστε σήμερα εδώ στην Επιτροπή μας. Ένα από τα θέματα τα οποία δεν αναφέρατε εσείς είναι το θέμα της εγγύησης για τα παιδιά. Στην 3 Δεκεμβρίου συμφώνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα επόμενα του Προσεγούς Κοινωνικού Ταμείου να, γίνει, ε, να υπάρξει ένα κονδύλι περίπου 6 ε, δις για να καταπολεμηθεί η φτώχεια των παιδιών. Πράγμα το οποίο θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα παρά το γεγονό ότι υπήρχαν ενδιασμοί εκ μέρου τη Επιτροπή, η Ισπανική κυβέρνηση και η κυρία Φάντερ Λέιν είπαν απερίφραστα ότι θα πρέπει να υπάρχει κοινωνική πολιτική για τέτοια θέματα που πιστεύαμε ότι πλέον έχουν εκριζωθεί από τις κοινωνίες μας. Και αναφέρομαι ειδικά στο θέμα αυτό της φτώχειας των αυτών. Πιστεύουμε ε, ότι Τέτοιου είδου όμως δεσμεύσει δεν θα πρέπει να προσέχονται από κονδύλια μόνο του Κοινωνικού Ταμείου συν, αλλά να υπάρχει μια ειδική πρωτοβουλία ώστε να υπάρχει συγχρηματοδότηση και διαχείριση των κονδυλίων αυτών για να μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική. Η Ευρώπη των ε, ε, ευκαιριών, κύριε Κούρτσε, αρχίζει από την παιδική ηλικία. Και θα πρέπει να απαντήσετε στο ερώτημα γιατί υπάρχει τέτοιου τους καθαστέρηση. Τι πιστεύετε ότι θα μπορείτε να μας ε, προσφέρετε τώρα που επομίστηκε αυτή την ε, πρωτοβουλία και η νέα ε, πρόεδρος της Επιτροπής. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς ώστε να μην ε, αποδυναμωθεί ακόμη μία φορά το θέμα αυτό. Κυρία Φράντση, ευχαριστώ Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Κόρτ για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Έχω δύο σύντομα ερωτήσεις, αλλά συγκεκριμένες. Πώς εκτιμάτε την εργασία που κάνουν οι Ευρωπαϊκές Επιτροπές Επιχείρησης και τι έχετε να πείτε εσείς για το θέμα της μετάθεσης κάποιων εργαζομένων ε, και για ανώτατο όριο 5 ετών. Πώς αποτιμάτε το θέμα αυτό. Τελευταία ερώτηση τώρα. Ήταν αυτή και έχει τον λόγο μέχρι τις 12 ε, παρατέρα του κύριο Κόρτσα για να απαντήσει. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις ε, ερωτήσεις που αφορούν πάρα πολλά θέματα και ίσως θα απογοητεύσω κάποιους από εσά, διότι σήμερα δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα κάνει η επόμενη Επιτροπή. Αλλά ε, κάποια θέματα θα τα απαντήσω. Για τον κύριο Ράτκε, ναι, ε, λέτε ότι στις εθνικές συζητήσεις ε, το κοινωνικό ζήτημα δεν παίζει σημαντικό ρόλο. Έχουμε το ίδιο πρόβλημα και παρόλο ε, που με τον πρόεδρο Γιούνκερ το έχουμε πει τόσες φορές δεν έχει επιτευχθεί η κοινωνική Ευρώπη να μπει κομμάτι της ε, εθνικής συζήτησης. Φαίνεται σαν δύο διαφορετικά επίπεδα που δεν συνδέονται μεταξύ τους. Ε, είναι δύσκολο και ανησυχητικό αυτό, όμως από την πλευρά της Κομισιόν θα κάνουμε ό,τι μπορούμε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων επικοινωνίας, ε, για να με τις ανακοινώσεις ε, μας ε, να το πετύχουμε αυτό. Επίσης, η ελάχιστη αμοιβή, συλλογικές διαπραγματεύσεις, όλα αυτά είναι αυτά που είπε και η κυρία Φόντερ Λάιεν. Είναι πολύ σημαντικά. Να, πού βρίσκομαι για να δω. Εδώ τις πρώτες 100 μέρες ε, της εντολής μου θα προτείνω ένα νομικό εργαλείο ώστε να διασφαλίσω ότι κάθε εργαζόμενος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα δίκαιο ελάχιστο μισθό. Αυτό θα σημαίνει ότι θα ζουν αξιοπρεπώς. Οι ελάχιστες αμοιβέ θα πρέπει να ορίζονται βάσει των εθνικών ε, παραδόσεων μέσα από συλλογικές διαδικασίες ή ε, δίκες ε, διατάξεις. Ε, πιστεύω στον κοινωνικό διάλογο και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις οι άνθρωποι που γνωρίζουν τον κλάδο ξέρουν καλύτερα. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Είτε θα έχουμε ελάχιστο μισθό μέσα από την νομοθεσία, είτε μέσα από τον κοινωνικό διάλογο. Παρεμπιπτόντας, όταν μιλάμε με τους νομομαθείς μας για τις δυνατότητες που υπάρχουν σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο που διέπει αυτή την επιλογή, ε, δεν μπορούμε να πάρουμε αυτή τη δικαιοδοσία από τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ένα πολύ θεμελιώδες στοιχείο και δεν έχει και νόημα. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν θέλουμε να εξασθενήσουμε τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις, αν υπάρχουν ακόμα καλύτερα. Αλλά αν υπάρχει τρύπα, ε, όπως υπάρχει στην Σουηδία ή ακόμα και στη Δανία, καλό είναι να γίνει αυτή η συζήτηση. Κύριε Γιονκέρες, ε, ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας, οι πολιτικές ε, δεσμεύσεις θα είναι εκεί δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα τι θα γίνει. Ξέρω όμως ότι το θέμα ανεβαίνει στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε ήδη φτιάξει μια ομάδα στο μικρό μας κόσμο της Επιτροπής που συνδυάζει όλες τις υπηρεσίες ε, που εμπλέκονται. Μιλάμε για θέματα όπως τις ευκαιρίες ε, που έχουν τα κράτη-μέλη για να δώσουν κρατικές χορηγήσεις έχουμε τους συναδέλφους από την Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, π.χ., για να βρουν μια στρατηγική που θα αντιμετωπίσει ακριβώς αυτές τις αυξανόμενες απαιτήσεις στην κοινωνία μας. Όταν μιλάμε τώρα για την ε, οδηγία για την ε, οικονομία των πλατφορμών, η νέα πρόεδρος της Κομισιόν έχει σκοπό να εξετάσει αυτό το θέμα και από τη δική μας πλευρά νομίζω ότι έχει νόημα αυτό, όμως είμαι στα χέρια των πολιτικών ε, προϊσταμένων μου. Αν λένε στις ομιλίες τους ότι θα εξετάσουν τις συγκεκριμένες απαιτήσει που χρειάζονται για την οικονομία των πλατφορμών, όπως είπατε συγκεκριμένα και εσείς, ε, τα παραδοσιακά είτε για τους εργαζόμενους είτε για τους ε, εργοδότες, η συνθήκη μιλάει για εργαζόμενους, είναι σημαντικές, γιατί στα κράτη-μέλη ε, θα υπάρχουν τεράστιες επιπτώσεις στους μισθούς, στην κοινωνική ασφάλιση, στις συντάξεις. Και το θέμα αυτό φαίνεται ότι δεν είναι, είναι μάλλον άσχετο. Και αναρωτιόμαστε πώς θα αντιδράσουν τα κράτη-μέλη. Ο κύριος Κράτκε είπε πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα, πρέπει να γίνει μια ευρωπαϊκή συζήτηση γιατί δεν μπορείς απλώς να νομοθετείς σε μια χώρα και να νομίζεις ότι όλα είναι καλά. Υπάρχει η διασυνοριακή διάσταση, ε, υπάρχει η οδηγία για τις αποσπάσεις ε, η οποία ε, θα υποσκάψει το σύστημά σου. Κυρία Μπρουνέ. Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού αυτού κατοφλίου την έχουμε αναφέρει και στην παρουσίασή μου. Ε, μιλάμε για την οικολογική επίσης μεταμόρφωση. Και εδώ έχουμε ένα μεγάλο διακύβευμα. Για άλλη μια φορά, η νέα πρόεδρος της Κομισιόν είπε ενδιαφέροντα πράγματα, η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιοποίηση των κοινωνιών μας, ε, για αυτήν έχουν μεγάλη σημασία. Θα έχουν τεράστιες επιπτώσεις στον κόσμο της εργασίας και θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν πρωτοβουλίες για τον ελάχιστο μισθό. Έχω ήδη εκφραστεί. Κυρία Λάγκεν Ζίμπεν, εγώ δεν είμαι υπεύθυνο ε, για τον τομέα της υγείας. Όμως, Υπάρχουν ε, πολλές, ε, πολλοί τομείς όπου διασυνδέεται το δικό μου ας πούμε, χαρτοφυλάκιο με την υγεία. Στην ερώτησή σας μιλάτε για την νομοθεσία. Συμφωνώ μαζί σας. Ε, εντάξει, ε, με την νομοθεσία το, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δόντια για να δαγκώσει αν δεν ακολουθούν τα κράτη-μέλη. Αυτά που καλό θα ήταν να γίνουν. Όμως ε, για τον ελάχιστο μισθό έχω και μια απάντηση. Κυρία Ζουμέ, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Εργασίας Νομίζω ότι αυτό το γραφείο θα έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει σας συμβουλεύω να διαβάσετε τον ε, βασικό κανονισμό που αναφέρει ακριβώς ε, ποια είναι τα καθήκοντα αυτού του γραφείου που θα ε, ιδρυθεί στην Φλάβα και θα δείτε ότι βασικά θα επικεντρώνεται στην ευρωπαϊκή Ε, εργασία. Από το 1958 έχουμε φτιάξει ένα τεράστιο σώμα νομοθετικό. Ε, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, πολλά καλύπτονται ε, είτε από οδηγίε είτε από κανονισμούς, εξυγχρονίζουμε κατά διαστήματα, όμως αυτό που λείπει είναι κάτι που να μας προστατεύει από τις καταχρήσεις Εκεί πραγματικά ε, απογοητεύομαι ιδιαίτερα. Αν συγκρίνουμε τι γίνεται ας πούμε στον τομέα των τελωνίων, το ότι υπάρχει μια υπηρεσία τελωνίων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ την ίδια στιγμή για την επιθεώρηση εργασίας έχουμε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο, απογοητεύομαι. Είναι μια κουλτούρα. Είναι σημαντικό να φτιάξουμε μια κουλτούρα, να αυξηθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα ξεκινήσει αυτό το γραφείο. Μάλιστα το Διοικητικό Συμβούλιο στις 17 Οκτωβρίου θα συνέλθει για πρώτη φορά και ε, θα έχουμε και εκπρόσωπο ε, του Κοινοβουλίου για να μπορέσει να ε, συνεισφέρει και αυτό στο Διοικητικό Συμβούλιο. wage, Ελάχιστος μισθός. Νομίζω ότι και αυτό το κάλυψα. Πάντως πρέπει να σας πω, και ο κύριος Ντάνιελ το έθεσε αυτό, Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και οι δύο τις ιδιαιτερότητες του σκανδιναβικού μοντέλου. Το ζήτημα αυτό με έχει απασχολήσει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, τους 18 μήνες που είμαι στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και προερχόμενος από εκεί που προέρχομαι, μου κάνει εντύπωση αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχουν κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν διοργανώσει τα κοινωνικά του συστήματα με τρόπο καλύτερο από ό,τι δικές σας χώρες. Πολλοί φοβούνται ότι εξαιτία τη κοινοτική νομοθεσία, αν ένα κράτο μέλο φτάσει στο επίπεδο αυτό, θα έρθει η κοινοτική νομοθεσία έπειτα να αποδυναμώσει το σύστημα αυτό. Αυτό όμω δεν ισχύει στην πράξη και προκαλεί μια κάποια απογοήτευση, θα έλεγα. Νομίζω ότι θα πρέπει να διασκεδάσουμε τρόπον την, την ανησυχία αυτή, το φόβο αυτό, που θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ιδεολογικής φύσης δεν νομίζω ότι υφίστανται πραγματικά προβλήματα και δεν νομίζω ότι χώρες όπως οι δικές σας που έχουν βάλει τον πύχη πολύ πιο ψηλά από κάποιε άλλε χώρε σε ζητήματα όπω ο κατώτο μισθό, ουσιαστικά θα υπονομευτούν από την κοινοτική νομοθεσία. Οι συλλογικέ συμβάσει δεν διακυβεύονται σε καμία περίπτωση και σαφώ σέβεται το ζήτημα αυτό η κυρία Φοντελάιν, όπω είπε άλλωστε και στην αρχική τη εναρκτήρια ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Στεχόφσκι τώρα αναφέρθηκε στην ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Ξέρετε ότι είναι ένας από τους οργανισμούς μας που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της δικής μου γενικής διεύθυνσης. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος συμβάλλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη όλων αυτών των απαραίτητων δεξιοτήτων που απαιτούνται για όλους τους Ευρωπαίους. Μας βοηθάει ο οργανισμός αυτός να γνωρίζουμε ποιες είναι οι αναγκαίες απαιτούμενες δεξιότητες στην αγορά εργασίας. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το θέσω αυτό με καλύτερο τρόπο. Πάντως άκουσα κάποια επικριτικά σχόλια. Μπορούμε να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στο ζήτημα αυτό. Αναφερθήκατε εδώ πέρα στην βοήθεια προς τους νέους, τους ανήλικους στην Αυστρία. Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε εδώ πέρα σε συγκεκριμένους δείκτες επιδομάτων όσον αφορά τα ανήλικα παιδιά. Ουσιαστικά εδώ πέρα θέλουμε να καλύψουμε εργαζόμενους από την Τσεχία, την Σλοβακία, οι οποίοι εργάζονται στην Αυστρία και οι οποίοι δεν θα πρέπει βέβαια να λαμβάνουν, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή, χαμηλότερα επιδόματα τέκνων από αυτά τα οποία θα λάμβανε ένας Αυστριακός εργαζόμενος. Σαφώς θα πρέπει να διορθώσουμε την κατάσταση αυτήν. Κύριε Ντάνιελσον, θέσατε ένα συγκεκριμένο ερώτημα όσον αφορά την ασφάλεια στο χώρο εργασία. Όπως σα είπα τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε εισάγει ανώτατα επίπεδα για ορισμένες καρκινογόνες ουσίες. Μας είπατε ότι θέλετε να θέσουμε ένα στόχο μηδενικών εργατικών ατυχημάτων. Συμφωνώ με αυτό και πρέπει να δούμε βέβαια από κοινού αλλά και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς μπορούμε να προωθήσουμε ένα τέτοιο στόχο. Νομίζω ότι σαφώ θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με το ζήτημα αυτό και όντω νομίζω ότι δεν έχουμε επικεντρωθεί επαρκώ στο ζήτημα αυτό, τη καταπολέμηση δηλαδή εξάλληψη των εργατικών ατυχημάτων και θανάτων. Ο κύριο Μέντερ μα είπε ότι ανήκοντα ηλικιακά στου άνω των 50, μίλησε για του πιο ηλικιωμένου εργαζόμενου. Τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν εδώ πέρα ότι κινούμεθα στη σωστή κατεύθυνση. Το ποσοστό των ε, ανθρώπων που εργάζονται στην ηλικιακή αυτή ομάδα έχει αυξηθεί. Πάντως η ε, λεγόμενη αυτή ε, ασημένια οικονομία είναι απαραίτητη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να χρησιμοποιήσω μια ακόμα φράση που λέγεται συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρέπει κανείς να μείνει εκτός, δεν πρέπει κανείς να μείνει πίσω. Και για δεροντικούς και ηθικούς λόγους, αλλά και κυρίως επειδή δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή πλέον αν δείτε την κατάσταση της αγοράς εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έχει σήμερα, υπάρχει σαφής έλλειψη εργαζομένων σε πάρα πολλούς τομείς. Επομένως, το να μην χρησιμοποιούμε το εφιστάμενο εργατικό δυναμικό, το οποίο προέρχεται και από τους ηλικιωμένους ή το οποίο προέρχεται από τα άτομα με αναπηρία, είναι κάτι το απαράδεκτο. Προφανώς θα πρέπει να αξιοποιήσουμε επαγγελματικά και αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Νομίζω ότι πραγματικά χάνουμε όταν δεν το κάνουμε αυτό ένα σημαντικό ποσοστό του ανθρώπινου ενεργητικού κεφαλαίου. Και νομίζω ότι ε, όλα τα κράτη-μέλη, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τέτοια τα κράτη-μέλη θα θέλουν να δουν όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες να ενεργοποιούνται και να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά. Όσον αφορά μια επικείμενη νομοθεσία για την ε, ψηφιοποίηση, νομίζω ότι απάντησα στο ερώτημα αυτό. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις μικρές επιχειρήσεις, στις οποίες αναφερθήκατε, συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι η νέα πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις ε, ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις, τις οποίες δεν θα πρέπει να βαραίνει. Ένα πολύ σημαντικό άχθος. Ο κύριος Ματζορίνο αναφέρθηκε σε πολιτικές για τους ε, ηλικιωμένους, το κάλυψε αυτό, κάλυψε επίσης και το ζήτημα των πολιτικών για τους αστέγους, κάλυψε και το ζήτημα του κατώτου του μισθού. Κυρία Μπλικεμβιτσούτε, αναφερθήκατε εσείς στον κοινωνικό πυλώνα. Νομίζω ότι ε, το σχέδιο δράσης για τον κοινωνικό πυλώνα απαντά ουσιαστικά στο ερώτημά σα. Προφανώ παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στα όσα κάνουν τα κράτη-μέλη μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ξέρετε ότι για κάθε χώρα υπάρχουν συγκεκριμένε απαιτήσει οι οποίε απορρέουν από τον κοινωνικό πυλώνα. Και έπειτα έχουμε και τον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων, το scoreboard, όπου μπορούμε πραγματικά και να αξιολογήσουμε και να αποτιμήσουμε τι επιδόσει των επιμέρου κρατών μέλων. πάντω. το Ευρωπαϊκό Σχέδιο δράση μπορεί πραγματικά να μα βοηθήσει να κάνουμε έναν απολογισμό των δραστηριοτήτων που έχουν αναλυφθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση από όλα τα κράτη-μέλη. Πρέπει να δούμε να ακολουθούνται συγκεκριμένε αρχέ, ποιε είναι οι μονομένε δράσεις των κρατών μελών και να δούμε και το ζήτημα τη διακυβέρνηση του πυλώνα, πώς οργανώνται τα κράτη-μέλη προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ο πυλώνας Όντω εφαρμόζεται στην πράξη. Στη δική σας τη χώρα, για παράδειγμα, τη Λιθουανία, έχουν δοθεί κάποια πολύ θετικά παραδείγματα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη υπηρεσία της κυβέρνησής, αν δεν κάνω λάθος, που ασχολείται με την επιτήρηση εφαρμογής του κοινωνικού πυλώνα σε όλα τα Υπουργεία. Τώρα, ελάχιστο εισόδημα, το οποίο δεν είναι το ίδιο με τον κατώτατο μισθό βέβαια, και Γι' αυτό προσπαθούμε να δούμε τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να κάνουμε μια απογραφή δηλαδή της κατάστασης και έχουμε συστήσει και μια ομάδα μελέτη στην οποία συμμετέχουν τα κράτη-μέλη, η εργασία της οποίας ακόμα είναι σε εξέλιξη και ελπίζουμε ότι θα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα με την νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Γερμανική Προεδρία, η οποία θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμεινο του επόμενου έτους, θα επιληφθεί του ζητήματος αυτού και νομίζω ότι με το ζήτημα αυτό έχει ήδη ασχοληθεί και η γερμανική κυβέρνηση. Νομίζω λοιπόν ότι ήδη υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ήδη έχουν αναλυφθεί δράσει. Δεν ξέρω αν θα αναλάβει συγκεκριμένε δράσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τώρα τι εγγύσει για τα παιδιά. Η κυρία Τζινέλα αλλά και άλλοι συνάδελφοι μίλησαν για το ζήτημα αυτό. Πάλι το μόνο μπορώ να κάνω να αφαιρθώ στο λόγο τη νεοκλεγή σα Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ανέλαβε συγκεκριμένε δεσμεύσει όσον αφορά τα επιδόματα τέκνων, είπε ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν όλα τα παιδιά και γι' αυτόν το λόγο θα δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά βασιζόμενη σε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λέει η νεοκλεγή πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μέσω του εργαλείου αυτού κάθε παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένο ή στο περιθώριο από κοινωνική πλευρά θα έχει πρόσβαση σε κατάρτιση και σε κοινωνικά προγράμματα. Θα δοθούν πολλά εκατομμύρια ευρώ, όχι αστείευουμε αυτό, δεν το ανέφερε, δεν αποτίμησε ακριβώς τα κονδύλια τα οποία θα δοθούν, αυτό απομένει ακόμα να το δούμε. Και κάτι το οποίο θα μπορούσα να αποτολμήσω να πω αυτή τη στιγμή αυτή είναι ότι δεν είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει να αναγκάσουμε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά να συμβάλλει χρηματοδοτικά στο κονδύλιο αυτό για την εγγύηση για τα παιδιά, γιατί ορισμένα κράτη-μέλη έχουν μικρή συμμετοχή ή πολλές φορές έχουν άλλες προτεραιότητες. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να εξατομικεύσουμε λίγο την κατάσταση και η πρωτοβουλία αυτή να εφαρμοστεί περισσότερο εκεί που πραγματικά υφίσταται η ανάγκη. Πάντω, νομίζω ότι αυτό θα το εξετάσουμε λίγο περισσότερο σε επικείμενου τριμερεί διαλόγου. Όσον αφορά τι τις, επιτροπές εργαζομένων, έχουμε δημοσιεύσει ένα ενημερωτικό φυλάδιο και προσπαθούμε να δούμε με τους κοινωνικούς εταίρους αν θέλουν να προχωρήσουν λίγο περισσότερο, πέρα δηλαδή από την υφιστάμενη συμφωνία που υπάρχει. Αυτή τη στιγμή όμως εργοδότες και εργαζόμενοι δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν μια κάποια συμφωνία για το τι θα μπορούσε να διαδεχθεί την οδηγία αυτή για τις επιτροπές εργαζομένων. Χρειαζόμαστε πάνω στη δική του συμβουλή για να προχωρήσουμε περισσότερο. Όσον αφορά την απόσπαση των εργαζομένων, υφίσταται μια έκθεση την οποία επεξεργάζεται η φυστάμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή της υφιστάμενης οδηγίας. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για τη νέα οδηγία. Πρέπει να παρακολουθήσουμε περισσότερο την εφαρμογή της υφιστάμενης οδηγίας και τον Μάιο του 2020 θα μας σε να υποβάλουμε μια νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως εμείς αυτή τη στιγμή ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζουμε νέους κανόνες, νέες ε, κατευθυντήρες γραμμές όσον αφορά τους νέους κανόνες απόσπαση. Το κείμενο είναι ήδη διαθέσιμο και μεταφράζεται αυτή τη στιγμή σε επίσημες γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ήδη υπάρχει μια ομάδα κρατών μελών που πιλωτικά μας βοηθά για να αποτιμήσουμε σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς εφαρμόζονται στην πράξη οι νέοι αυτοί κανόνες για την απόσπαση των εργαζομένων. Πολύ εργασία όμως ακόμα πρέπει να γίνει του επόμενου μήνε και τα επόμενα χρόνια για το ζήτημα αυτό. Σας ε, ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετική εργασία επιτελέσετε προσπαθώντας να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Με εντυπωσιάσατε. Είναι ακριβώς 11.47 στα χρονικά μας πλαίσια. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση, για τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των συναδέλφων και προσβλέπουμε σε περαιτέρω συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ. So, συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε με την παρουσίαση μίας μελέτης Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΟΕ, διαμορφώνοντας το μέλλον το εργασιακό. Θα ήθελα να δώσω πρώτα απ' όλα το λόγο στον συντάκτη της έκθεσης αυτής, τον καθηγητή Φραντσέσκο Παστόρο. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να παρουσιάσω την uh, μελέτη αυτή. Νομίζω ότι η μελέτη αυτή είναι πάρα πολύ χρήσιμη, διότι θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τη σχέση που υφίσταται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που είναι ένας από τους βασικούς, αν θέλετε, καθοριστικούς παράγοντες ε, στο διεθνές προσκήνιο, ιδίως στον τομέα των κοινωνικών προβλημάτων και κυρίως της αγοράς εργασίας. Θα μιλήσουμε λοιπόν και αν μπορούμε να περάσουμε και στην επόμενη διαφάνεια. για τη διαρθρωτική σχέση που υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΔΟΕ. Ας δούμε λίγο και τη δομή της μελέτης αυτής. Ένα τμήμα της μελέτης έχει να κάνει με το μέλλον της εργασίας. Θα ήθελα επίσης να σας κάνω μια σύντομη ιστορική αναδρομή της σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και για κάθε μία από την περίοδο αυτή που έχουμε εντοπίσει θα σας δίνω και το γενικότερο ιστορικό πλαίσιο, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Στο τελευταίο τμήμα της παρουσίασης, που είναι και το τελευταίο τμήμα της μελέτης, θα αναφερθούμε στο ίδιο το μέλλον της εργασίας, δηλαδή νέα βιομηχανική επανάσταση, νέα βιομηχανική εξέλιξη, η λεγόμενη βιομηχανία 4.0, όπως θα δείτε, λέμε ουσιαστικά ότι η εξέλιξη αυτή είναι λιγότερο δραματική από ό,τι προτείνουν κάποιες άλλες μελέτες. Λοιπόν, μια αρχική αιτιολόγηση για τη μελέτη αυτή. Για ποιο λόγο είναι η μελέτη αυτή. Θεωρήσαμε ότι ήταν θετικό το ότι συμπίπτει χρονικά με την εκατοστή επέτειο του Διεθνούς Γραφείου Συνεργασίας και με την 60η επέτειο της Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΔΟΕ. Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε όταν θεσπίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και ουσιαστικά η τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ένα χρόνο δηλαδή μετά την υπογραφή της συνθήκης της Ρώμης, θα δείτε ότι η αρχική αυτή περίοδος ήταν μια περίοδος άτυπης συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών αυτών. Έκτοτε όμως η συνεργασία αυτή ήταν πάρα πολύ σημαντική για να καθοριστεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και νομίζω ότι ε, τα τελευταία αυτά 60 χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια συγκεκριμένα, όπως άλλωστε δείχνει και η μελέτη μας, η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Γραφείου Εργασίας βασίζεται ουσιαστικά σε αυτή την κοινή εργασία που έγινε από τους δύο οργανισμούς, σε αυτές τις πολύ συστηματικές συναντήσεις, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο της έντονης προσπάθειας που κατέβαλαν και οι δύο οργανισμοί. Νομίζω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει να έχουμε και μία εναλλακτική, αν θέλετε, επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι βασίζονται στη συνθήκη του Μάστριχτ, προκειμένου να επικεντρωθούν περισσότερο σε ένα σημαντικό επίτευγμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που σύμφωνα με αυτού είναι το Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη, εμεί βασιζόμενοι στη συνεργασία με το Διεθνέ Γραφείο Εργασία, θα θέλαμε να τονίσουμε αν θέλετε του κοινωνικού στόχου που έθεσε τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να δημιουργήσει ένα πιο θετικό πλαίσιο απασχόληση, προκειμένου να θέσει επαγγελματικού και κοινωνικού στόχου. Και νομίζω ότι στόχος της μελέτης αυτής είναι να εξετάσει λίγο περισσότερο πώς φτάσαμε, αν θέλετε, στους στόχους αυτούς μέσω της συνεργασίας που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Να πω και λίγα λόγια για τη μεθοδολογία την οποία ακολουθήσαμε, καθώς επίσης και τις διαθέσιμες πηγές. Πρόκειται για την πρώτη μελέτη η οποία έλαβε χώρα για τη συνεργασία αυτή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Είχαμε κάποιες ε, πρωταρχικές και δευτερογενείς πηγές. Χρειάστηκε να εξετάσουμε τα πρακτικά των ε, συνεδριάσεων υψηλού επίπεδου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Συνεδριάσεις οι οποίες έλαβαν χώρα προκειμένου να υπάρχει σύγκληση απόψεων μεταξύ των δύο οργανισμών για τα σημαντικά κοινωνικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν την εποχή εκείνη. Έπειτα καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή με κάποιους προνομιούχους συνομιλητές οι οποίοι ήταν κέρι, αν θέλετε, παράγοντες στη συνεργασία αυτή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΔΟΕ και καταφέραμε κατά αυτόν τον τρόπο να αποσπάσουμε και να αντλήσουμε πληροφορίες οι οποίες πουθενά αλλού δεν ήταν διαθέσιμες. Γι' αυτόν τον λόγο καταλήξαμε σε μία καινοτόμα μελέτη με στοιχεία τα οποία ουδέποτε έχουν συλλεχθεί και ουδέποτε έχουν παραχθεί και εκτεθεί κατά αυτόν τον τρόπο στο παρελθόν. Νομίζω ότι η μελέτη αυτή τονίζει όλο και περισσότερο τη σημασία και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Από μεθοδολογικής πλευράς θα ήθελα να σας πω ότι για κάθε κεφάλαιο έχουμε μία συγκεκριμένη ανάλυση, θεωρητική καταρχάς, δηλαδή μια γενική συζήτηση της πολιτικής που ακολουθείται, των βασικών εκτιμήσεων, των βασικών συζητήσεων του Παλαβανχώρα χώρα και στη συνέχεια προσπαθούμε μέσω της μελέτης να δείξουμε πώς οι θεωρητικές αυτές ιδέες γίνανε συγκεκριμένη πολιτική, γίνανε συγκεκριμένες δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια τα περισσότερα έγγραφα τα οποία χρησιμοποίησαμε ως πηγές είναι τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο τμήμα της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ξεκίνησε το 1958. Στην αρχή η συνεργασία αυτή είχε τη μορφή άτυπων συναντήσεων και η σχέση μεταξύ των δύο οργανισμών ήταν περισσότερο η σχέση που έχει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν εξωτερικό οργανισμό. Την εποχή εκείνη η Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρωνόταν πολύ περισσότερο σε εσωτερικές της εξελίξεις, επομένως αρχίσανε να γίνονται λίγο περισσότερο, αν θέλετε, διεθνείς παίκτες ε, οι Ευρωπαίοι όσον αφορά τον απτυσσόμενο κόσμο, από θεωρητική όμω πλευρά, γιατί δεν είχαν ούτε την απαραίτητη γνώση, αλλά ούτε τα απαραίτητα κονδύλια ή του απαραίτητου οικονομικού πόρου, προκειμένου να βοηθήσουν ε, τρίτε συναπτυσσόμενε χώρε. Γι' αυτό το λόγο την εποχή εκείνη η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ιδίω στο πλαίσιο των εξωτερικών υποθέσεων και της εξωτερικής συναπτυξιακής βοήθειας βασιζόταν στην εμπειρογνωμοσύνη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας προκειμένου να βοηθήσει τις συναπτυσσόμενες χώρες. Όπως θα δείτε και στην επόμενη διαφάνεια, μια σειρά συναντήσεων έλαβαν χώρα, αρχικά άτυπες συναντήσεις, οι οποίες γινόντουσαν όλο και πιο επίσημες, συναντήσεις που γίνανε μεταξύ λοιπόν των δύο αυτών οργανισμών και στις οποίες είχαμε όλο και περισσότερο παρατηρητές και από τις δύο πλευρές. Μέσω των άτυπων αυτών συναντήσεων έγινε μία μηδέ προσπάθεια κατανόησης του ενός οργανισμού από τον άλλον, χωρίς όμως να υπάρχουν ακόμα επίσημες μέθοδοι συνεργασίας. Τα πρώτα έγγραφα στα οποία μπορούμε να δούμε την επίδραση τη θετική του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας είναι η Λευκή Βίβλος την οποία συνέταξε ο Ζακ Καντελόρ όσον αφορά τις κοινωνικές πτυχές στις πολιτικές που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδίως στον τομέα των επενδύσεων και της οικονομικής ανάπτυξης. Από το έγγραφο λοιπόν αυτό μπορούμε να δούμε πιο ξεκάθαρα την επιρροή, τη θετική επίδραση της συνεργασίας με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Δεν θα επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τη διαφάνεια αυτή. Προς ενημέρωσή σας απλώς σας τις δείχνω. Καταγράφεται εδώ πέρα η όλη εργασία την οποία κάναμε προκειμένου να εχνηλατήσουμε τα διάφορα βήματα της εξελισσόμενης εργασίας, συνεργασίας μάλλον, μεταξύ των δύο αυτών οργανισμών. Βλέπετε πόσο πιο έντονη γινόταν η συνεργασία αυτή, προϊόντος του χρόνου, πως σιγά σιγά πέρασαν από πιο άτυπες μορφές συνεργασίας σε πιο επίσημες μορφές συνεργασίας. Έπειτα έχουμε την άλλη περίοδο, από το 2000 έως το 2007, περίοδο κατά την οποία το Διεθνές Γραφείο Εργασίας άρχισε να συνεργάζεται πιο συστηματικά και πιο επίσημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συναντήσεις υψηλού επίπεδου αρχίσαν να γίνονται όλο και πιο συχνές και συστηματικές μεταξύ των ανώτατων αξιωματούχων των δύο οργανισμών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη μια πλευρά, Διεθνές Γραφείο Εργασίας από την άλλη. Υπάρχει μια σημαντική συνάντηση μεταξύ του τότε, διεθνούς, μεταξύ του τότε Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και του τότε Επικεφαλής Ευρωπαϊκής Επιτροπής του κυρίου Ρωμάνο Πρόντι και βλέπουμε ότι υπάρχει και μια πιο έντονη και επίσημη συνεργασία μεταξύ μονομένων επιτρόπων και ανώτων αξιωματούχων από το διεθνέ Γραφείο Εργασία, Από τα πρακτικά των συνεδριάσεων και των συναντήσεων αυτών μπορούμε να δούμε και κάποια ιστορικά ορόσημα, Σημαντικέ συνεδριάσει που έλαβαν χώρα και σημαντικέ αποφάσει που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων αυτών προκειμένου να καταφέρουμε ήδη από τότε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες κοινωνικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το ακολουθηταίο κοινωνικό μοντέλο. Την περίοδο μάλιστα αυτή από το 2000 έως το 2007 δηλαδή έχουμε και μια όλο και μεγαλύτερη συμβολή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να εγκαθιδρυθεί μια πιο βιώσιμη συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών. Σε σχετικές εκθέσεις και πρακτικά μπορείτε να δείτε λεπτομερέστατε συζητήσει για όλα τα ζητήματα τα οποία απασχολούσαν τότε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νέες θέσεις απασχόλησης, φιλοπεραβολαντικές θέσεις απασχόλησης κ.ο.κ. Θεωρώ ότι μελετώντα κανεί τα κείμενα αυτά μπορεί να συνειδητοποιήσει πόσο πολύ είχε προχωρήσει τότε και σε τι βάθος είχε προχωρήσει τότε η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Θεωρώ λοιπόν ότι πραγματικά αξίζει να διαβάσετε τις σχετικές αυτές εκθέσεις αλλά και τη μελέτη μας, καθώς επίσης και τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων από τους δύο αυτούς οργανισμούς. Εμείς μέσω της μελέτης μας προσπαθήσαμε να σας δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες σε χρονολογική σειρά όσον αφορά τις συναντήσεις αυτές που έλαβαν χώρα την περίοδο 2000 με 2007. Τώρα, το 2007 είχαμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα σε συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών. Όπως ξέρετε, ξέσπασε τότε η οικονομική κρίση και η σχετική συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών άρα ασχολείται περισσότερο με τις δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης και ιδίως με την ανεργία και την ενεργία των νέων. Ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αυτό που πρώτο πρότεινε την πρωτοβουλία για τους νέους, το Youth Guarantee, και από τη μελέτη μας όμως μπορούμε να δούμε ότι το ζήτημα αυτό είχε απασχολήσει και τους συμμετέχοντες στις συναντήσεις με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας έχοντας τη θετική εμπειρία των σκανδιναβικών χωρών ήταν και αυτό σε θέση να προτείνει πρωτοβουλίες παρεμφερείς με το Youth Guarantee, με την πρωτοβουλία απασχόληση των νέων, που όπω είπε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε πρώτο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε αυτήν και σε επόμενες διαφάνειες βλέπετε ότι η μελέτη μας επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στο ζήτημα του μέλλοντος της εργασίας. Η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Γραφείου Εργασίας άρχισε με την πάροδο του χρόνου να επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στο νέο αναδυόμενο εργασιακό περιβάλλον. Περάσαμε όλο και περισσότερο από μέτρα αντιμετώπιση τη ανεργία και δι τη ανεργία των νέων προ συζητήσει οι οποίε αντιμετώπιζαν με μεγαλύτερη ισοδοξία πλέον τι μελλοντικέ μορφέ εργασία και συζητήσει οι οποίε θέλουν να αναδείξουν τον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι πολίτε θα μπορούσαν να αποφεληθούν από τι νέε μορφέ εργασία προκύπτουν, αλλά και από φαινόμενα όπω η αυτοματοποίηση ή η ψηφιοποίηση της εργασίας. Προσπαθούμε εδώ πέρα να βασιστούμε στις θετικές εμπειρίες κρατών μελών και προσπαθούμε να διασκεδάσουμε τρόπον την και εμεί τις ιδιαίτερα καταστροφικές προβλέψεις που κάνουν κάποιες άλλες μελέτες οι οποίες μιλούν για μια ευρεία μαζική καταστροφή πολλών θέσεων απασχόλησης όπως τις γνωρίζουμε σήμερα. Εμείς στη δική μας μελέτη αναφερόμαστε σε μια σειρά από μελέτες όπως η μελέτη Frey Osborne του 2015 που λέει ότι ένα 47% των θέσεων απασχόλησης πρόκειται να καταργηθούν μέσω της νέας αυτής μορφής εργασίας. Από την άλλη υπάρχουν άλλες μελέτες οι οποίες προτείνουν σχετικά ποσοστά τα οποία είναι πολύ πιο χαμηλά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ο πρώτος περιορισμός σε αυτή τη μελέτη και η διαδοχικές ε, μελέτες δείχνουν ότι μάλλον όλες οι δουλειές θα αλλάξουν σύν το χρόνο ως ε, επίπτωση ας πούμε, της αλλαγής ε, του τρόπου εργασίας, όμως λίγες θα καταστραφούν. Φαίνεται ότι μόνο στο 10% θα είναι σε αυτή την κατηγορία και αυτό είναι κι άλλος ένας περιορισμός των μελετών γιατί κοιτούν μόνο την καταστροφή των θέσεων εργασίας. Όμως αυτή η επανάσταση δημιουργεί και θέσεις εργασίας. Έχουμε νέες δουλειές, η καινοτομία θα μειώσει το κόστος της εργασίας. Αυτό θα επιτρέψει νέες παραγωγές να είναι εφικτές και οικονομικά δυνατές. Άρα, εκτός από την καταστροφή των θέσεων εργασίας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε στη μελέτη είναι να επικεντρωθούμε στις επιπτώσεις των πολιτικών, στα επίπεδα των πολιτικών όμως, καλό είναι όταν κοιτάμε τις μελέτες του ILO και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βλέπουμε και πώς λειτουργεί η καινοτομία. Οι επενδύσεις στην καινοτομία μας βοηθάνε να περάσουμε πιο γρήγορα στο στάδιο της δημιουργίας θέσεων εργασίας και να φύγουμε από το στάδιο της καταστροφής. Αυτό είναι λοιπόν ο στόχος μας, να προχωρήσουμε να αυξήσουμε την καινοτομία, την ταχύτητα της καινοτομίας για να φτάσουμε στο στάδιο της δημιουργίας θέσεων εργασίας και να γίνει αυτό πιο γρήγορα. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό τομέα ε, μοντέλο είναι το καλύτερο ε, που ε, θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Ε, για να αντιμετωπίσουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Και για να ολοκληρώσω ε, στον χρόνο μου να πω ότι προσπάθησα να συνοψίσω το περιεχόμενο της μελέτης όσο πιο καλά μπορούσα. Να καταλήξω λοιπόν με ένα τομέα με μια πτυχή που είναι πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μας. Ο κοινωνικός διάλογος είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία της ανάλυσης της σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εθνούς Γραφείου Εργασίας. Λαμβάνουν αποφάσεις μεν, αλλά διευκολύνουν και την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. Αυτό είναι το σημαντικό στη συνεργασία τους. Και κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι οι πηγές δεν είναι αρκετές. Θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα στοιχεία. Για να ολοκληρώσω την ομιλία μου, να πω ότι στις χώρες, στα κράτη-μέλη δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση για τη σημασία αυτής της συζήτησης. Μιλάμε συνήθως για το μέλλον της εργασίας, δεν ξέρουμε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν ήδη συντάξει προτάσεις, έχουν θεσπίσει πολιτικές που θα μειώσουν τους κινδύνους και θα αυξήσουν τις ευκαιρίες. Άρα προτείνω όχι μόνο να δείξουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα θέματα, αλλά να προσπαθήσουμε να τις προβάλλουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης περισσότερο, διότι είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε και αυτή την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο της χρηματοπιστωτικής και νομισματικής σταθερότητας. Νομίζω ότι το ευρωπαϊκό εξάμεινο για τα κοινωνικά ζητήματα θα μπορέσει να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον ε, καθηγητή Παστόρε και τώρα δίνω το λόγο στην ε, κυρία Φερπόβεν. Σας καλωσορίζω. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, εξότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε ως Διευθύντρια του ΑΕΛΟ στο Γραφείο των Βρυξελών, που συνδιαλέγεται με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Μετά από την παρουσίαση της μελέτης για τα 60 χρόνια συνεργασίας μεταξύ Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η σημερινή συνάντηση είναι επίκαιρη. Γιατί, Γιατί ξεκινά μια νέα θητεία στην ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολύ σημαντικό για μας, αλλά επίσης επειδή φέτος ε, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας ε, γιορτάζουμε τα 100 χρόνια μας. Η ιστορία του ILO είναι μεγαλύτερη από αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ε, υπάρχουν και πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ των δύο ιστοριών. Ο ILO ε, δημιουργήθηκε με τη συνθήκη των Βερσαλιών μετά από έναν ε, πόλεμο που κατασπάρεξε όλη την Ευρώπη. Έτσι, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας κατάφερε να εφαρμόσει μια παγκόσμια κοινωνική ειρήνη ε, αυτό που ήταν και η καρδιά της θητείας του. Έχουμε λοιπόν μια εταιρική σχέση όχι μόνο με τα κράτη αλλά και με τις οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων. Αργότερα μετά από άλλη μία καταστροφική σύραξη η Ευρώπη επανενώθηκε ε, βάσει των ίδιων ιδεών της ίδιας λογικής. Ο κοινωνικός διάλογος λοιπόν είναι στο DNA του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και του μοντέλου του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Γιατί σας θυμίζω το Ρεζόν Τέτρε, το λόγο ε, δημιουργίας και ύπαρξής μας. Ε, γιατί είναι σημαντικό επειδή τώρα ως θεσμοί αντιμετωπίζουμε προκλήσεις στην αγορά εργασίας και πάντοτε πρέπει να σκεφτόμαστε τις ρίζες μας από όπου ξεκινήσαμε. Οι κοινέ αξίες που έχουμε, οι δεσμεύσει μας το αποδεικνύουν. Κοιτάξτε για παράδειγμα το επίπεδο κύρασης των βασικών στάνταρ προτύπων εργασιακών προτύπων. Ε, και τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ε, κυρώσει αυτές τις διεθνείς ε, συμβάσεις, εργασιακές συμβάσεις που οι κυβερνήσεις, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι των 187 κρατών μελών μας έχουν συμφωνήσει και θεσπίσει. Αφού κυρωθούν αυτά, γίνονται νομικά δεσμευτικά έγγραφα και στη συνέχεια εφαρμόζονται διεθνώς στα μέλη του ILO. Δεν έχουμε μόνο νομοθεσία, έχουμε και συστάσεις για εργαλεία, πολιτικές, βέλτιστες πρακτικές που προωθούν οι συστάσεις και οι συμβάσεις. Τώρα, λίγα λόγια για την συνεργασία, ε, για να συμπληρώσω τη μελέτη. Μετά από 60 χρόνια συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμών, μπορώ να πω ότι έχουμε όλο και μεγαλύτερη, όλο και πιο ευρεία, εντατική και βαθιά συνεργασία. Γιατί είναι πιο ευρεία. Η μελέτη δείχνει ακριβώς μια σειρά επιλεγμένων θεμάτων επί των οποίων συνεργαζόμαστε. Όμως υπάρχει και η μετανάστευση, η παγκόσμια λυσίδα τροφοδοσίας. Ε, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν αυξήσει το μέγεθος της μελέτης. Αν δεν υπήρχαν θα ήταν μισό το μέγεθός της. Όπως είπε και ο καθηγητής, έχουμε τις συναντήσεις υψηλού επίπεδου, έχουμε πιο ε, τακτικές συναντήσεις που είναι σε επίπεδο επικεφαλής του ILO και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε τις γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά έχουμε και από τον ILO ε, ανθρώπους οι οποίοι συνεργάζονται με DG, DG Trade, DG Mare, DG AFCO, με όλες αυτές τις διευθύνσεις όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και με άλλα θεσμικά όργανα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή σας ε, τακτικά, με άλλες επιτροπές, την ΙΝΤΑ, ΦΑΜ, ΔΕΒΕ, ΛΥΜΠΕ. Υπάρχουν και άλλα ε, θεσμικά όργανα με τα οποία συνεργαζόμαστε, όπως ο πούμε και επίσης ε, τα γραφεία, υπάρχει μία ad hoc ομάδα συμβουλευτική η οποία ας πούμε περιλαμβάνει τον ILO ως εμπειρογνώμονα, ε, ως παρατηρητή. Αυτό είναι ένα πολύ απτό παράδειγμα της πιο εντατικής και ευρείας συνεργασίας μας. Και τέλος να πω ε, ότι τα τελευταία αυτά 60 χρόνια υπήρξε μια εμβάθυνση αν ε, δείτε ακριβώς τι, έχουν γίνει αυτά τα, τι έχει γίνει αυτά τα 60 χρόνια, υπήρξε όλο και περισσότερη τεχνική συνεργασία. Το Κοινοβούλιο ανοίγεται προς άλλες ε, χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το νούμερο ένα τα τελευταία 10 χρόνια ως ε, δωρητής μέσα στα πλαίσια της τεχνικής συνεργασίας με τον ILO. Επίσης έχουμε 7 συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου ε, που μας επιτάσσουν να εφαρμόζουμε συγκεκριμένα στάνταρτ ελεύθερου εμπορίου. Όλα αυτά είναι στην καρδιά των διαπραγματεύσεων και υπήρχαν, υπήρξαν και εργαλεία για τον ILO για να προωθήσει τα στάνταρτ στον χώρο της εργασίας, τα βασικά στάνταρτ που αφορούν δηλαδή την παιδική εργασία, την αναγκαστική εργασία, τις ίσες ευκαιρίες, τις μη διακρίσεις και τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις. Αυτή η συνεργασία είναι πολύ σημαντική για τον ILO και μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αλλά και σε διεθνές επίπεδο π.χ. στο G20 και σε άλλους σχηματισμούς είμαστε έτοιμοι να δράσουμε. Όλα αυτά τα θέματα ε, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε άμεσα. Έχουμε τον οδικό χάρτη με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Χρειάζεται πλήρης εφαρμογή. Ο ΕΛΟ έχει επιμεληθεί του κειμένου και στα επόμενα χρόνια ε, ελπίζουμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Θέλουμε λοιπόν στη διακήρυξη των 100 ετών να μιλήσουμε για αυτούς τους στόχους και να συνεργαστούμε περαιτέρω, να αλλάξουν τα πράγματα για τους ανθρώπους, για τον κόσμο της εργασίας. Τέλος, αυτό που θα ήθελα να κάνω δράτοντας την ευκαιρία σήμερα, καθώς συνεχίζουμε τη συνεργασία μας, είναι να σας δείξω κάποιους συγκεκριμένους τρόπους ε, συνεργασίας, α, ας πούμε. Που θα είναι χρήσιμα και για σας και για τους βοηθούς σας. Τι κάναμε στο παρελθόν μοιραστήκαμε όλες τις στατιστικές, τις πληροφορίες, τα στοιχεία που είχαμε ε, από το σύστημα εποπτείας των στάνταρ των εργασιακών. Κάναμε διάφορες ενημερωτικές συνεδριάσεις με εισηγητές, συνεισηγητές, briefing ε, πριν να πάνε αντιπροσωπείες σε διάφορες χώρες στα πλαίσια του Διεθνούς Οργανισμού και Είπαμε πώς χρησιμοποιούνται τα εργασιακά στάνταρ στην νομοθεσία και σε άλλα επίσημα έγγραφα. Τα... Εξηγήσαμε όλες αυτές τις δυνατότητες που υπάρχουν. Συμπερασματικά, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η συνογραφία μεταξύ των δύο οργανισμών μας σε αξιοπρεπή εργασία και σε κοινωνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο είναι επίκαιρο και απαραίτητο και για την Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Ευχαριστώ και είμαι έτοιμη να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δύο προσκεκλημένους μας για την ε, ομιλίες τους. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στους συντονιστές. Ο κύριος Ράτκια, εκ μέρους του ΕΛΚ. Δεν τον βλέπω όμως. Εκ μέρους των σοσιαλιστών, η κυρία Ιαχαρίς. Ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε πολύ για τις μελέτες, για την παρουσίαση και για το ότι εξετάζετε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και στα πλαίσια της Επιτροπής αλλά γενικότερα και από όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σας. Όντως, από την προηγούμενη εργασία μου έχω κάποια εμπειρία από το Διεθνές Γραφείο Εργασίες το οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα. Και τις ε, κηρύξεις που έγιναν στα πλαίσια του διάσκεψης του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας στα πλαίσια του ε, μέλλοντος για την εργασία και βλέπω ότι στα πλαίσια αυτής της εργασίας λαμβάνονται υπόψη όλοι οι εταίροι. Υπάρχουν νέοι τομείς εργασίας, δεδομένου ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες που ανοίγονται εξαιτία της ψηφιοποίησης και αυτό οδηγεί στο να υπάρχουν πολλοί αυτοαπασχολούμενοι και δημόσιοι φορείς, κυβερνήσεις που πρέπει να μοιράζονται ψηφιοποιημένες πλατφόρμες και να δουλεύουν με νέους τρόπους. Μπορεί κανείς να εργάζεται και από τις διακοπές του. Στα πλαίσια των ε, μελετών σας προβλέπετε στα πλαίσια αυτών των νέων μορφών ψηφιοποιημένης εργασίας να συζητήσετε κάποια εξελίξεις, κάποιες νέες προτάσεις στα πλαίσια όλων όσων ενέχονται σε αυτές τις νέες μορφές εργασίας, εργοδότες και εργαζόμενους. Ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω ότι έχετε παρακαλώ δύο λεπτά κάθε συνάδελφος για να Έχουμε χρόνο. Κύριος Πισλάρου, ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για τα εκατοστή επέτειό σας στο Άγιελου. Εξ ονόματος του Renew θα πρέπει να πω ότι σας συγχαίρω το έγγραφό σας, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο και μπορεί να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε περαιτέρω λήψη αποφάσεων. Εμείς θα θέλαμε να έχουμε μία σύγχρονη Ευρώπη που να έχει ισχυρό κοινωνικό και οικονομικό σχέλος και νομοθεσία που να είναι σωστή και για τους εργοδότες και για τους εργαζόμενους. Κυρίως στα πλαίσια της διαμόρφωσης της εργασίας στο μέλλον είχαμε πάρα πολλά ερωτηματικά και πολλά έχουν ε, λεχθεί πώς θα γίνουν τα πράγματα, υπάρχουν απογοητεύσει, υπάρχουν ερωτηματικά. Το πρόβλημα δεν είναι απλώς να επιβιώσουμε. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε να γίνουν τα πράγματα και να επιβιώσουμε. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση εμείς να οδηγήσουμε κατά κάποιο τρόπο τις εξελίξεις και να προβλέψουμε πώς θα δημορφούν τα πράγματα και έχουμε λοιπόν μία πρώτη σειρά πολιτικών που οδήγησαν σε στάνταρ, σε ισότητα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτή την αδέση. Αλλά το δεύτερο στάδιο είναι να σκεφτούμε, να εστιάσουμε στο μέλλον, ώστε να μπορέσουμε στα πλαίσια μιας νέας στρατηγικής και εφιού στρατηγικής να προλάβουμε κάποια γεγονότα για να ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Η ερώτηση είναι, μπορεί να μας εξηγήσετε τι σκέφτεστε για θέματα που απασχολούν τις κοινωνίες μας, όπως ε, η κυκλική οικονομία, η μετανάστευση, ε, νέες μοφές εργασία, δημιουργία ε, νέων θέσεων εργασίας, τα πλαίσια της ψηφιοποίησης, πλατφόρμες, πράσινες θέσεις απασχόλησης. Θα πρέπει, όπως σας είπα, να είμαστε ένα βήμα, ένα κλικ μπροστά από τα γεγονότα. Ευχαριστώ. Η κυρία Πίτερ Χάνσον, εκ μέρους των Δεν είναι παρούσα. Η κυρία Λάγκε Ζίπμεν επίσης δεν είναι εδώ. Η κυρία Ζαμέ δεν είναι επίσης παρούσα, εκ μέρους της ID. Από την ECR, η κυρία Ραφόλσκα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα Στο πλαίσιο της ε, συνεργασίας αυτής των 60 ετών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, σαφώς ε, μας ενδιαφέρει πολύ η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, αλλά πολλά πράγματα, πολλά διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε και από την ίδια την ιστορία. Μπορούμε με βάση τη ιστορική αυτή συναδρομή να δούμε ακριβώ πώ θα διαμορφωθεί στο μέλλον η συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών και ιδίω όσον αφορά το λεγόμενο μέλλον τη εργασία. Αναφερόμαστε όλο και περισσότερο σε ζητήματα ψηφιοποίηση. Η πρόεδρο λέει ότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα με τη διερμηνία. Till then. So you have your two minutes, you can start again. Please. Ας περιμένουμε λιγάκι, θα αποκατασταθεί το πρόβλημα. Έχω μία ερώτηση. Δεδομένου στι νέε τεχνολογίε πρέπει να βλέπουμε και τι νέε ευκαιρίε που ανοίγονται. Ποιοι είναι όμω οι κίνδυνοι που επίση θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια τη υγείας, της ψυχολογικής κατάστασης, της οικογένειακής κατάσταση του καθένα, Λαμβάνεται υπόψη διάφορου κινδύνου, οι οποίοι ενέχονται και όχι μόνο τις ευκαιρίες που ανοίγονται. Εκ μέρους της Γκουέ, η κυρία Χάιμπη. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για αυτή την πλήρη παρουσίαση. Επιμένετε πολύ στο πόσο σημαντικός είναι ο κοινωνικός διάλογος. Και είπα, ναι, επαναλαμβάνω αυτά που είπατε, ότι ο κοινωνικός διάλογος ήταν μέλος του DNA στα πλαίσια των κοινωνικών σχέσεων. Στην, ένα, στην ε, σελίδα 106 μιλάτε για το γεγονός ότι πρέπει να ανανεώσουμε, να δώσουμε, προσδώσουμε μια νέα σημασία στον κοινωνικό διάλογο και υπάρχει ε, στα πλαίσια των συλλογικών ε, διαπραγματεύσεων στην Ευρώπη και του κοινωνικού διαλόγου μια επιδείνωση. Δεν μας εξηγείτε για ποιες Ποιοι είναι οι λόγοι του οποίου υπάρχει επιδείνωση, παρά το γεγονό ότι εξηγείται ότι είναι πάρα κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη δημοκρατία. Ποια είναι η άποψή σα, δεδομένου ότι στην έκθεση αυτή υπάρχει η διασύνδεση μεταξύ Διεθνού Γραφείου Εργασία και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των πολιτικών ε, ε, λιτότητας που προβλέπονται στα πλαίσια το Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των πρόσχερων και επισφαλών συνθηκών εργασίας και της μείωσης της ισχύς της ε, συλλογικής διαπραγμάτευσης. Επίσης κάπου αλλού λέτε ότι η οικονομία στις πλατφόρμες συνεισφέρει στην επιδείνωση του κοινωνικού διαλόγου. Εξηγείται το εξή. Οι εργαζόμενες πλατφόρμες δεν είναι μισθωτοί. Και λέτε σωστά ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε τις νέες μορφές οργάνωσης των εργαζομένων ή αυτοοργάνωσης των εργαζομένων. Υπάρχουν πολύ μεγάλες κινητοποίησεις παντού στην Ευρώπη, κυρίως στη Γαλλία, με τα εργαζόμενους της υπηρεσίας delivery, στον delivery όπως λέει στη Γαλλία. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, ίσα δικαιώματα κοινωνικά και ασφαλιστικά για να μπορέσουν να έχουν και εκείνη τη σύνθεση εργασία με τους άλλους εργαζόμενους. Ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο σε άλλους συναδέλφους, αν θέλουν να κάνουν ερωτήσεις ή παρατηρήσεις. Εάν κάποιος όντως θέλει το λόγο, να σηκώσει το χέρι του τώρα. Δεν βλέπω κανένα συνάδελφο, άρα θα δώσω το λόγο στους ε, προσκεκλημένους μας, πρώτα απ' όλα στον κύριο καθηγητή, για να απαντήσει. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλες οι ερωτήσεις είναι ενδιαφέρουσες και πραγματικά αξίζει να απαντηθούν. Η πρώτη ήταν ε, για τους ε, εργοδότες. Είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να υπάρξουν να υπάρξει μεγαλύτερη εμπλοκή των ε, εργοδοτών γιατί οι εργοδότες είναι οι βασικοί παράγοντες αν θέλουμε να εφαρμόσουμε τις νέες τεχνολογίες. Είναι σημαντικό οι εργοδότες να καταλάβουν πως ο ρόλος τους δεν είναι μόνο να παράγουν. Πρέπει ας πούμε να δώσουν κάποια κάποιες χορηγήσεις στους νέους ε, για να μπορούν ε, να ε, αντιμετωπιστούν, να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες. Η αρχή του διτού συστήματος, του εκπαιδευτικού συστήματος, όχι μόνο πανεπιστήμιο, αλλά και βιομηχανικά PhD, βάσει αυτού του συστήματος. Αυτό το σύστημα θα είναι ο οδηγός, ας πούμε, για την μετατροπή του συστήματος, την ε, συγχώνευση. Ένα άλλο θέμα είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι μόνο χώρος παραγωγής ή κατάρτισης, αλλά και χώρος καινοτομίας. Θα πρέπει να καινοτομούν περισσότερο οι επιχειρήσεις. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να τονίσουμε είναι το εξής. Επειδή είναι πολλές ερωτήσεις θα προσπαθήσω να απαντήσω έτσι κάπως σύντομα. Οι επιχειρήσεις ε, διαθέτουν σημαντική γνώση για την επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα είναι σημαντικό κεφάλαιο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Νομίζω ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να το συνειδητοποιήσουν αυτό. Πρέπει να τις πιέσουμε να καινοτομήσουν περισσότερο, να αναπτύξουν καινοτομία ως προς τις πολιτικές για το μέλλον της εργασίας. Αναφέρθηκε ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες πολιτικές, για χάρη συντομίας ανέφερα μερικές. Η προστασία της ποιότητας της εργασίας είναι επίσης σημαντική. Αν την προστατέψουμε, θα οδηγήσουμε τις εταιρείες, τις επιχειρήσεις προς την καινοτομία, προς εργασίες υψηλής ποιότητας για να μειώνεται το εργασιακό κόστος ε, και να μην ε, διαλύεται, ας πούμε, ε, να μην υπάρχει διάλυση των θετικών στοιχείων της καινοτομίας. Δυστυχώς η διερμηνία θα σταματήσει λόγω λήξης της βάρδιας μας. Last question. Uh, the uh, platform work was also uh, uh is, uh, is dealt in details in, in the study